Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της σημερινής τη σημερινή συνεδρίαση μάλλον. Si se van sentando, por favor. Καθίστε σας παρακαλώ. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της συνεδριάσεως είναι η έγκριση των πρακτικών του σχεδίου της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε σχόλια και δεν έχετε προσθήκες, μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Καλώς, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχουμε τίποτα σε αυτό το σημείο. Α, κάτι έχουμε. Ε, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Νατσόνη θα... Η κυρία Ματσόνη θα προείδρευε, δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει το πρωί, θα έρθει, θα έρθει αργότερα και έτσι έχω εγώ την τιμή επειδή και πρώτος και δεύτερος αντιπρόεδρος δεν είναι εδώ, εγώ έχω την τιμή να προεδρεύσω σαν τρίτος αντιπρόεδρος στα διάφορα θέλετε να θέσετε κάποιο θέμα. Όχι. Οπότε πάμε στο σημείο 5 της... Μάλλον ανακοινώσεις του Προέδρου πάμε τώρα, τις αποφάσεις των συντονιστών, συνεδρίασαν το πρωί οι συντονιστές. και συζήτησαν το, τα θέματα που είχαν στη μερίσια τους διάταξη. Να σας πω ότι αποφασίστηκε για να ξέρετε πρώτα-πρώτα συζητήσαμε όσον αφορά την ακρόαση που θα γίνει το 2011 στην Επιτροπή μας και όπως ξέρετε την τελευταία συνάντηση οι συντονιστές, όχι σήμερα, στην προηγούμενη, αποφασίσαμε να γίνει μια κρόση όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών για τις αναφορές και αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι στην επόμενη συνέντευξη όλο αυτό να συζητηθεί Δεύτερο σημείο που συζητήθηκε είναι το τι θα γίνει με τις μη αναφορές, γιατί όπως γνωρίζετε είχαμε συζητήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες ή μήνες τι θα γίνει με τις μη αναφορές. Με ό,τι δεν αναφορά τέλο πάντων και αποφασίστηκε η διοίκηση να το μελετήσει και να μας πει οι δύο γενικητές το συζητούν τώρα και θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία τις αμέσως επόμενες μέρες. Οπότε, θα περιμένουμε την επιστολή του Γενικού Διευθυντή για να το συζητήσουμε. Και όταν λάβουμε αυτή την επιστολή, θα προχωρήσουμε στο σημείο τώρα υπαριθμών 3. Είπαμε τι θα γίνει με την νομοθεσία για τις ακτές. Και εδώ είπαμε να γίνει μια συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές και τους, αναφε, ε, τους πάντων, και ζητήθηκε μια γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας, η οποία από την νομική υπηρεσία πριν από λίγες μέρες μας στείλανε στα αγγλικά μια γνωμοδοτηση νομική υπηρεσιας η οποια απο υπηρεσια πριν Είπαμε να μεταφραστεί και περιμένουμε τη μετάφραση. Σήμερα περιμέναμε να έχει φτάσει η μετάφραση, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πάμε επομένω στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Φαντάζομαι τότε θα έχουμε τη μετάφραση. Ο κύριος Βοστινάρου ζήτησε στη συνάντηση του Δεκεμβρίου να μιλήσουμε για τα μέσα ενημέρωση στη Ρουμανία. Είπαμε να περιμένουμε μέχρι ότου μιλήσουμε του αρμοδίου. Συμφωνώ και ο Και βέβαια θα καλέσουμε επομένω όταν έρθει η ώρα και τι ρωμανικέ αρχέ και του αναφέροντε Να έρθουν εδώ στη συνεδρίαση. Αυτά αποφασίστηκαν από του συντονιστέ. Pregunta sobre, la reunión de coordinadores. Θα έπρεπε να αναφέρετε την απόφαση για την admin. Με va a έχετε δίκιο. Και μου είπε η κυρία Οκέν ότι δεν είδα την πίσω σελίδα όπου αναφέρεται η τελευταία απάντηση, η τελευταία απόφαση των συντονιστών. Εκεί λέμε ότι θα πρέπει σε μια ε, μελλοντική συνάντηση Τι, τι είναι κυρία Άκυν, τι είπαμε. Α, ήταν το θέμα που αφορά τις σχέσεις Ισραήλ-Ένωσης. Συμπαθάτε με που δεν είδα την πίσω σελίδα. Θα συντηθεί στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα τη ημέρα διάταξη. Ο λόγο θα δοθεί στην κυρία Wallis. Έχουμε και την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά μια πρωτοβουλία των πολιτών. Κυρία Γουόλης, έχει το λόγο για το σχετικό νομοθέτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνήσαμε ο κ. Χάφνερ να αναφερθεί στο θέμα. Ο κ. Χάφνερ, λοιπόν, έχει το λόγο. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Η Νταϊάννα Βόλης και εγώ συνεργαστήκαμε. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά, συγκεντρωμένοι αυτό το μήνα επί της εκθέσεως και συνεργαστήκαμε με δύο εισηγητές της ΑΦΚΟ, Ζήτα Γκόμαε και τον κύριο Λαμασούρ. Αυτό που μπορούμε να προτείνουμε σήμερα είναι ένα σχέδιο κανονισμού όπου έχουμε συμφωνήσει σχεδόν επί όλων των σημείων. Υπάρχουν μικροδιαφορές που απομένουν μεταξύ του δικού μας σχεδίου εκθέσεως, υπάρχουν διαφορές, και αυτού που συζητείτε στην ΑΦΚΟ. Την ίδια μέρα συζητείτε το θέμα στις δύο επιτροπές. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι στο τέλος να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκφράζεται σε μια έκθεση που θα υποβληθεί ταυτόχρονα από την ΑΦΚΟ και την Επιτροπή Αναφορών. Αν τα καταφέρουμε να το κάνουμε, θα ληφθεί τελευταία απόφαση από αυτού στην Σύνοδο του Δεκεμβρίου στο Στασβούργο. Πριν από αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε το σχέδιο εκθέσεως. Το προτείνουμε σήμερα και θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση η κυρία Βόλης και εγώ σας παρακαλούμε αν έχετε τροπολογίες ή προτάσεις να τις υποβάλλετε ούτω ώστε να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις μας και στην απόφασή μας στην επόμενη συνεδρίαση. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στα σημαντικότερα σημεία. Καταρχάς να πω ότι νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή αυτή για το Κοινοβούλιο και ειδικά για την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Αναφορών, διότι τώρα θα εισαγάγουμε ένα νέο μέσο για την συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα μέσο που θα επιτρέπει στους πολίτες άμεσα να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις. Δεν είναι ένα μέσο άμεσης δημοκρατίας. Δεν είναι μέσο λήψεως αποφάσεων και θέσπισης νομοθεσίας είναι ένα μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας και καθορισμού ημερησίων διατάξεων και προγραμμάτων, ε, ένα μέσο μέσω των οποίων μπορούν να υποβάλουν προτάσεις οι πολίτες. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει, εάν δημιουργηθεί σωστά και αν λειτουργήσει σωστά, είναι να δημιουργήσει πλαίσιο διαλόγου, ε, να υπάρχει διάλογος μεταξύ θεσμικών οργάνων και πολιτών. Και μέσω του διαλόγου θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια ενωμένη Ευρώπη, Ευρώπη των πολιτών, όπου θα έχει την εντύπωση ο πολίτη ότι εισακούγεται όταν έχει ανησυχίε ή προτάσει, ότι θα εισακούγεται τα θεσμικά όργανα, κυρίω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το μόνο θεσμικό όργανο που επιτρέπεται να υποβάλει προτάσει για νομοθεσία. Για να φτάσουμε εκεί όμω, είναι πολύ σημαντικό ο ίδιο ο κανονισμό να δημιουργεί το διάλογο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε πολλά μέτρα διατάξεις με τις οποίες θα πρέπει συμμορφώνονται οι πολίτες. Δεν αρκεί όμως αυτό. Θα πρέπει οι διατάξεις να εφαρμόζονται και από τα θεσμικά όργανα. Να ακούνε προσεκτικά δηλαδή τα θεσμικά όργανα τις επιθυμίες των πολιτών. Η μεγαλύτερη αποτυχία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μέσο να πούμε στον κόσμο ότι μπορείτε να υποβάλλετε προτάσεις και στο τέλος να τους δώσουμε την εντύπωση ότι κανείς δεν ακούει αυτά που θέλουν. Τώρα θα έρθω στα σημαντικότερα σημεία κατά την άποψή μας. Ξεκινήσαμε με το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Μαρτίου του 2010 και προσπαθήσαμε να κάνουμε το κείμενο λιγότερο γραφειοκρατικό, πιο φιλικό για τον πολίτη. Προσπαθήσαμε να διοργανώσουμε τον κανονισμό ε, με έναν τρόπο που πραγματικά να βοηθήσει τη δημιουργία αυτού του διαλόγου. Το θέμα ήταν της ε, καταγραφής, καταχώρησης και του, της αποδοχής. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρία στάδια. Αφού ξεκινήσει η πρωτοβουλία των πολιτών και αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνεται μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο καταγράφεται, καταχωρείται αυτό το αίτημα, αυτή η πρωτοβουλία και Επόμενο βήμα, αφού συλλεχθούν 300.000 υπογραφές, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει ένας έλεγχος νομικός για το αποδεκτό του αιτήματο και μετά αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια ή όχι. Νομίζουμε ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό αυτό. Είναι πολύ γραφειοκρατικό να σταματήσει κάτι μετά από 300.000 υπογραφές όταν συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών και συνεχίζεται η εκστρατεία. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτό να το θέσουμε σε δύο σημεία, να το αναφέρουμε. Στην αρχή πρέπει να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο καλύπτεται, είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επιτρέπεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση επί του συγκεκριμένου ζητήματο, αν δεν είναι προφανώ κάτι που στρέφεται κατά των αξιών τη Ενώσεω, που αναφέρονται στο άρθρο 2 τη συνθήκη, των συνθήκων μάλλον, δεν δημιουργεί προβλήματα γέννη, δεν είναι κάτι γελίο, και αν όχι αρχίζει η συλλογή υπογραφών και δεν χρειάζεται να διακόψουν μετά από 300.000 υπογραφές. Για να μην υπάρξει πρόβλημα να αντιμετωπίσει εκατοντάδες ε, πρωτοβουλίες πολιτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά, προτείναμε να υπάρχει ένα πρώτο εμπόδιο. Δηλαδή, η πρωτοβουλία των πολιτών θα πρέπει να υποβάλλεται από μια επιτροπή οργανωτών Επτά άνθρωποι από επτά κράτη-μέλη πρέπει να είναι. Δηλαδή, ήδη έχει γίνει κάποια συζήτηση για το θέμα, το σκεφτήκαν διεξοδικά, το προετοίμασαν και είναι ικανοί να διοργανώσουν τη συλλογή των υπογραφών. Αυτό θα μας βοηθήσει να ε, υποβάλλονται πιο σοβαρές προτάσεις και να αποφύγουμε το εμπόδιο των 300.000 υπογραφών. Τώρα, ποιος επιτρέπεται να υπογράψει δεν είναι απαραίτητο αυτό να συσχετιστεί με το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές. Δεν είναι ψήφος, δεν είναι λήψη απόφασης, δεν είναι αισμευτική απόφαση, είναι απλώς προτάσεις και θέλουμε και οι νέοι να μπορούν να το κάνουν. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει αναφορά και έτοιμα παρά την ηλικία του ή της. Δεν υπάρχει όριο για την πρωτοβουλία των πολιτών, προτείνουμε την ηλικία των 16 για να επιτρέψουμε και στου νέου να υποβάλουν προτάσει. Όσον αφορά τον αριθμό των κρατών μελών, προτείνουμε το 1 πέμπτον των κρατών μελών και όσον αφορά το θέμα του πώς γίνεται επαλήθευση των υπογραφών, λέμε ότι δεν είναι θέμα ταυτοποίησης του κάθε μέλους, εκεί θα είχαμε πρόβλημα όσον αφορά τους νόμους για την προστασία των δεδομένων, αλλά θα πρέπει να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να δούμε κατά πόσο αυτοί που γράφουν είναι πολίτες, κατά πόσο έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν και αν υπέγραψαν μία φορά. Για να μην υπάρχουν διπλές υπογραφές και ονόματα. Και να παραμείνει η διαδικασία απλή και έρχομαι σε κάτι σημαντικό στο τέλος. Δεν ανεφέρω όλα τα σημεία, αλλά η Ντάνα Wallis και ο Ζήτα Κόμαε που είναι εδώ σήμερα, συζητή από την ΑΦΚΟ μαζί με τον Αλέα Λαμασούρ, μπορούν να συνεχίσουν. Για να μην χρησιμοποιήσω εγώ όλο το χρόνο. Τελευταίο σημαντικότατο σημείο κατά την απόψη μας είναι το εξή. Τι θα συμβεί αν έχουν συλλεχθεί από τους πολίτες ένα εκατομμύριο υπογραφές. Λέμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να παραμείνει κάτι ανοιχτό. Δεν θα αρκεί να πούμε στον κόσμο μέσω επιστολής ευχαριστούμε που συλλέξατε τις υπογραφές, δεν θα ακολουθήσουμε την πρότασή σας. Ε, πρέπει αυτή η τεράστια δουλειά που έχουν κάνει οι πολίτες να εκτιμηθεί από τα θεσμικά όργανα. Τι σημαίνει αυτό ότι πρέπει τουλάχιστον να διεξαχθεί μια ακρόαση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει τον κόσμο και να ακούσει τι προτάσει του τα επιχειρήματά του σε μια δημόσια ακρόαση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας, διότι στην κοινωνία των πολιτών όλοι μα ρωτούν γιατί να συλλέξουμε ένα εκατομμύριο υπογραφέ, τι θα συμβεί στο τέλο. Και το σχέδιο κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ασαφέ και ανοιχτό επ' αυτού και θέλουμε σαφή κανονισμό που θα λέει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να διεξαχθεί στο τέλος μία ακρόαση. Σας ευχαριστώ και προσβλέπουμε στις συζητήσεις και στις τροπολογίες σας, αν έχετε τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω μήπως θέλει το λόγο τώρα ή μετά. Κύριε Βόλης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπε ο κ. Χάφνερ για την καλή συνεργασία που είχαμε, εμείς οι τέσσερις συζητήτες. πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος μέσω συνδυασμένης προσέγγισης. Το έγγραφο που έχει μπροστά της η Επιτροπή διαφέρει ελάχιστα από αυτό της ΑΦΚΟ, αλλά σε αρκετά τα σημαντικά σημεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτα απ' όλα, η εμπειρία μας αφορούσε αναφορές που δεν υπήρχε λόγος για τις αναφορές αυτές να υπάρχει ένα κατώτερο όριο ηλικίας και θα έπρεπε να συμμετέχουν οι νέοι, να πνεύσουμε τους νέους να συμμετάσχουν στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Αυτή ήταν η εμπειρία μας εδώ στην Επιτροπή και αυτό θα θέλαμε να δούμε όσον αφορά το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Αυτό δεν είναι δικαίωμα ψήφου, είναι δικαίωμα υπογραφής μιας πρωτοβουλίας, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο να μην ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των νέων Νομίζουμε ότι θα ήταν ενδεδειγμένο αυτή η Επιτροπή με την ιστορία της, όσον αφορά τις αναφορές, να συνεχίσει να υποστηρίζει την αλόγω αρχή. Άλλη σημαντική πτυχή για την Επιτροπή μας αφορά αυτό που αναφέρθηκε. Δηλαδή, τι συμβαίνει μετά όσον αφορά την ε, επιτυχή πρωτοβουλία διότι πάνω απ' όλα εδώ χρειάζεται απόλυτη σαφήνεια. Δηλαδή εκείνοι που επιτυχώς συνέλεξαν το 1 εκατομμύριο υπογραφές, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις, τελικά να πετύχουν κάτι. Πολλοί από εμά θεωρούμε, και νομίζω κυρίως αυτή η Επιτροπή θα θεωρούσε, ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει κάποια θέση ή κάποια δυνατότητα να τοποθετηθεί όσον αφορά το μηχανισμό ανταπόκρισης και απάντησης. Σε πρώτη φάση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάτι στους πολίτες, γιατί είναι ο πρώτος παραλήπτης, ο πρωταρχικός παραλήπτης η Ευρωπαϊκή διότι ειναι ο πρωτος παραληπτης ο Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο αυτό το Κοινοβούλιο, όταν αυτό ενδείκνυται, δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται στη διοργάνωση κάποιας μορφής ακροάσεως ενδεχομένως σε κοινή συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για την Επιτροπή μας. Και θα ήταν ασυγχώρητο αν αυτή η Επιτροπή με την ιστορία της και την εμπειρία της δεν ε, προωθούσε αυτή τη δυνατότητα. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο διαφέρουμε ελαφρώς από τους συναδέλφους Επιτροπής ΑΦΚΟ. Πιστεύουμε ότι είναι μια απόκληση η οποία μπορεί τελικά να οδηγεί σε σύγκληση στο μέλλον. Διότι όλοι θέλουμε να πετύχουμε, πιστεύω, το καλύτερο δυνατόν για εκείνους οι οποίοι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να συλλέξουν αυτές τις υπογραφές. Υπάρχει και άλλο θέμα που αφορά το ποια θα είναι ανταπόκριση σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Πώς λειτουργεί, πώς αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες που θα έχει το Κοινοβούλιο όταν υποβάλει πρόταση ψηφίσματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς αντικατοπτρίζονται οι δύο διαδικασίες. Θα πρέπει παρομοίως να αντιμετωπιστούν τα δύο θέματα. Αυτές οι παράγραφοι χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, πιθανότατα περαιτέρω συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ειλικρινά Θέλω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Θέλω να ακούσω απόψεις και σκέψεις που θα μας δώσουν μια πλήρη εντολή. Πλήρη εντολή στην ομάδα των τεσσάρων εισηγητών για να προχωρήσουμε στις συζητήσεις με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Και βέβαια έχουμε και την προσδοκία να πετύχουμε συμφωνία πριν το τέλος του έτους για να διεξαχθεί τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αυτή όμως η προσδοκία δεν θα πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της σωστής λύσεως. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι το οποίο να είναι αντάξει όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προωθεί τη σχέση μας με τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Αγόλης. Στη συνέχεια δώσουμε το ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Όμως η συνάδελφο από την ΑΦΚΟ πρέπει να λάβει πρώτο λόγο ότι πρέπει να φύγει για να ψηφίσει η άλλη επιτροπή. Εάν δεν έχετε κάποια ένσταση, τότε να τη δώσουμε το λόγο. Κύριε Γκουρμάη. Ε, ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να σας μιλήσω σήμερα. Αυτό το θέμα της νέας πρωτοβουλίας πολιτών είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη στην Ευρώπη παντού μετά από την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η δική μας Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών και οι δύο γραμματείες βεβαίως μπόρεσαν να δουν ε, το θέμα αυτό με το, υπό το ίδιο πρίσμα και να επιτύχουν έναν υψηλό βαθμό συνένεσης. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να συγχαρώ την εξαιρετική εργασία της Κομισιόν διότι μας προσέφερε μια πάρα πολύ καλή βάση εργασίας. Ευχαριστώ τον ε, Μάριο, την Καμπριέλα, όλη την ομάδα. Χωρίς τη βοήθεια των πολύτιμων αυτών συνεργατών δεν θα είχαμε προχωρήσει ε, τόσο επιτυχώς. Η Βελγική Προεδρία και η Τρόικα των Προεδριών, Ισπανική, Βελγική και Ουγγρική, θεωρεί το θέμα αυτό υψής σημασίας. Με ένα πάρα πολύ καλό, με ένα εξαιρετικό έγγραφο εργασίας ε, κατά την Ισπανική Προεδρία μπορέσαμε και προχωρήσαμε έτσι επιτυχώς και γρήγορα. Η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών θα γίνει ένα βοήθημα στους Ευρωπαίους πολίτες για το πώς θα κατανοήσουν και θα δράσουν καλύτερα ως Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό κάθε φορά που δίνουμε ένα νέο δημοκρατικό μέσο στα, στα χέρια των πολιτών πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι τι θα συμβεί τώρα στην πρακτική, διότι αυτό εδώ είναι παρθένο έδαφος και δεν έχει ξαναγίνει. Σωστό ότι μετά από τρία χρόνια πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του μέσου αυτού. Πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει και με μια δημόσια ακρόαση, ποιο θα τη χειριστεί, πώς θα προχωρήσει η Κομισιόν, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα να σα θυμίσω ότι το άρθρο 11, παράγραφος 4 τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν λέει πάρα πολλά επ' αυτού, γι' αυτό ακριβώς και εμεί έχουμε μια ευχέρεια ε, χειρισμού της πρωτοβουλίας αυτής. Έχουμε ένα κοινό στόχο, ότι πρέπει να είναι επικεντρωμένο στους πολίτες, ότι βεβαίως οι, οι, οι παραχωρήσεις, τα δικαιώματα συνδέονται με καθήκοντα και υποχρεώσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει πρωταρχικό ρόλο να παίξουν τα ευρωπαϊκά θέματα, διότι αν τελικά καταλήξουμε να έχουμε 7 άτομα από 7 χώρες, αυτό θα είναι μια πάρα πολύ καλή κατάληξη. Και βεβαίω τα ουγγρικά χρειάζονται να μεταφραστούν τα κείμενα, αλλά βεβαίως όσο το δυνατόν περισσότερε ευρωπαϊκέ γλώσσε. Ε, Σα είπα ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και συζήτηση με τα στελέχη της Κομισιόν. Επίση, είναι σημαντικό να εγγυηθούμε ότι σεβόμαστε τι ε, οδηγίε και τι διατάξει τη Ευρωπαϊκή ε, Προστασία Δεδομένων ε, και ότι θα εφαρμόσουμε ένα δίκτυο εποπτείας για να δούμε αν τηρούνται τα κριτήρια. Ε, έπρεπε να είμαστε ρεαλιστές ε, κατά τη διαδικασία για να μπορέσουμε να αγγιηθούμε το καλύτερο δυνατόν εργαλείο μέσων αυτό που θα προσφέρουμε στους πολίτες μας. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα προχωρήσει υπό την Προεδρία του κυρίου Κασίνη στην Επιτροπή μας. Ε, συνεισηγητής μου ήταν ο κύριος Λαμασούρ, άλλος θαυμάσιος συνεργάτης και τον ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ε, ε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για έναν κοινό στόχο. Ας δούμε εάν μπορούμε να επιτύχουμε μια πρώτη ανάγνωση ή όχι. Όμως, χρειαζόμαστε μια πάρα πολύ καλή ποιοτική βάση ε, συνενετική και αυτό το έχουμε επιτύχει. Όπως πάντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα έχεις να μας πεις. Συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Τερνέιρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς τους δύο εισηγητές της Επιτροπής Αναφορών και της ΑΦΚΟ. Ήταν μία από τις πιο ολοκληρωμένες διαδικασίες και ικανοποιητικές τις οποίες μπορέσαμε να υποστηρίξουμε. Είχαμε και την κάλυψη του Συμβουλίου, άρα λοιπόν η θέση μας είναι ε, πολύ αισιόδοξη και επικοδομητική. Ελπίζουμε ότι σύντομα συνενετικά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το ζήτημα. Ε, όσον αφορά τις ακροάσεις, τα είπατε αυτά, εγώ θα κάνω πέντε σύντομες παρατηρήσεις τις οποίες θέλω να προσέξετε. Μπορεί ενδεχομένω ένα από τα πέντε αυτά θέματα να δημιουργήσουν ε, κάποιες δυσκολίες. Το θέμα είναι εάν ε, το μπορέσουμε σωστά να χειριστούμε το θέμα του, του, του, αποδεκτού, του αποδέξιμου, ε, ποιο, ποια θα είναι κατάλληλα προς επιλογή, ποια όχι κλπ. Ε, γενικά βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Πέντε μικρές παρατηρήσεις, σύντομες παρατηρήσεις. Και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε ακόμα ερωτήσεις. Το πρώτο είναι η δημόσια κρόαση. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακρόαση από την Κομισιόν. Δεν θα είναι μόνο γραπτή διαδικασία και ανταλλαγή επιστολών. Η Κομισιόν οπωσδήποτε θα συναντήσει τους διοργανωτές και θα τους ακούσουμε. Αυτό το λέμε σαφώς. Τώρα άλλο ζήτημα το δικό μας και το άλλο ζήτημα η δημόσια ακρόαση με το κοινό. Ε, πιστεύω ότι η Κομισιόν, αλλά οπότε κατάλαβε και από εσά, από την κυρία Βόλης, πιστεύω ότι σε αυτή τη δημόσια ακρόαση δεν πρέπει να, να προεδρεύει η Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι ο, το φορέας αυτός που θα λαμβάνει τα μηνύματα. Πιστεύω ότι το ηγετικό ρόλο θα πρέπει να τον αναλάβει το Κοινοβούλιο ε, και να οργανώσει τη δημόσια ακρόαση ή δυνατόν στην αρχή της διαδικασίας για να μπορέσει να λάβει υπόψη της και η Κομισιόν τα συμπεράσματα. Και βεβαίως εμείς θα συνεργαστούμε και θα υπάρχει εκπροσώπη και δική μας στη δημόσια ακρόαση, αλλά ηγετικό ρόλο θα πρέπει να την οργανώσει και να προεδρεύει το Κοινοβούλιο. Ένα άλλο, το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να θίξω, που ακόμα δεν έχει λυθεί τελείως, είναι η τροπολογία 46. Ο παραλληλισμός μεταξύ της πρωτοβουλίας πολιτών και της, ε, του, του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου επί του άρθρου 2 έως 5. Βασικά, η συνθήκη δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ των δύο διαδικασιών. Η Κομισιόν θα ανταποκριθεί θετικά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έχει καμία επίπτωση στην πρωτοβουλία των πολιτών. Ε, και τα δύο καλύπτονται. Δεν θα πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να προχωρήσουμε υπερβολικά στενά στον παραλληλισμό αυτών των δύο διαδικασιών. Το, το τρίτο σημείο είναι το help desk είναι σαφές ότι η Κομισιόν όταν θα γίνει ακριβώς η εγγραφή ε, θα προσφέρει όλη της τη βοήθεια στους διοργανωτές, θα μιλήσει μαζί τους για την ενημέρωση και βοήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό άρθρο επί του θέματος αυτού. Η Κομισιόν υλοποιεί τους, ε, τις νομοθετικές διατάξεις και θα συζητήσουμε με το διοργανωτή, αλλά δεν νομίζω να πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο. Το τέταρτο είναι οι γλώσσες. Δύσκολο θέμα. Πρέπει να το απλουστεύσουμε. Η θέση της Κομισιόν είναι να είμαστε όσο δυνατόν πιο απλή. Στην αρχή να χρησιμοποιηθεί μία γλώσσα για την εγγραφή, μετά θα κάνουμε όλα τα, τους ελέγχους, όλα τα, τα checks που χρειάζονται σε μία γλώσσα, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε γρήγορα. Και μετά οι οργανωτές μπορούν να προσθέσουν και άλλες γλώσσες ή άλλες μεταφράσεις αν θέλετε στο αρχείο ε, και η Κομισιόν θα κάνει ένα γρήγορο έλεγχο να δούμε αν υπάρχει κανένα λάθος ή κάτι ασύμβατο, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα σε όλους τους ε, οργανωτές να κάνουν εγγραφές, να εγγραφούν με όλες τις γλώσσες της κοινότητας, διότι θα δημιουργηθεί μια βαβυλωνία γλωσσών, ε, θα καθυστερήσει τις διαδικασίες και θα πρέπει να γίνουν ε, ε, ε, ενδελεχείς έλεγχοι μεταξύ των μεταφράσεων, αν είναι ακριβείς κλπ. Μεγάλη δηλαδή γραφειοκρατική καθυστέρηση. Και το πέμπτο σημείο οφείλεται σε μία πιστεύω παρανόηση. Είναι οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές τι εννοώ για τους Α, για το σύστημα συλλογής των υπογραφών online. Αυτή η διαδικασία θα είναι απλουστευμένη έτσι κι η Κομισιόν θα προσφέρει το λογισμικό, το software που μπορεί να χρησιμοποιήσει, το εγκεκριμένο, οπότε αυτό ήδη βοηθάει. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ε, η νομική βάση για τη συλλογή αυτή των ε, υπογραφών ε, υπάρχει ήδη στον κανονισμό, άρθρο 6.4. Δεν χρειάζεται τώρα να αναπτύξουμε τη νομική βάση για τις υπογραφές. Απλώς να βοηθήσουμε την ε, τεχνική διεκπαιρέωση αυτής της διαδικασίας. Σας είπα ότι ο κανονισμός ήδη καλύπτει, προσφέρει τη νομική βάση για τη συλλογή υπογραφών online ε, και είμαστε καλυμμένοι νομικά. Εάν λοιπόν υπάρχει παρανόηση, το διευκρινίζω. Αν θέλετε, έχετε καμία ακόμα απορία, απευθυνθείτε παρακαλώ σε μένα να σας το εξηγήσω. Ε, μπορεί βέβαια οι τεχνικές ε, προδιαγραφές ε, να δίδονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να υπάρχουν όλες αυτές οι υπογραφές. μέχρι ότου φτάσουμε στο σημείο όπου οι τεχνικές προδιαγραφές θα αποτελέσουν σώμα του, του νομοθετικού πλαισίου, θα είναι δηλαδή νομοθετικές. Αυτά ήθελα να πω. Είναι τα τελευταία πέντε ζητήματα που εκκρεμούν. Κύριε Τενέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και στη συνέχεια να δώσουμε το λόγο στην Προεδρία. Κύριε Χέρβαντ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε αυτή τη συνεδρίαση για αυτόν τον φάκελο, για αυτόν τον τοσχέ που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βελγική Προεδρία. Γι' αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το σχέδιο έκθεσης που, που μας προσφέρει ένα βήμα προόδου προς την υιοθέτηση αυτού του σημαντικού κανονισμού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές για την εργασία τους και τη θαυμάσια συνεργασία μέχρι τώρα στις, και όλους τους συνεργάτες της, ε, των ατύπων συνεδριάσεων που είχαμε με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Βεβαίως θα συζητήσουμε ε, τις ε, τροπολογίες το σχέδιο έκθεσης για να βρούμε τρόπους συμβιβασμού, και είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε πολλά, από τα δικά σας αιτήματα. Οι συζητήσεις δείχνουν ότι το Συμβούλιο θα σταθεί σε ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα, στα οποία ζητούμε την κατανόησή σας μέσα στο πνεύμα του συμβασμού. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά από αυτά τα ευαίσθητα σημεία. Ένα σημαντικό για το Συμβούλιο όπως ενδεχομένως θα έχετε ήδη διαβλέψει, είναι η διευκρίνηση των υπογραφών και το παράρτημα 3 του εγγράφου, το οποίο διαφέρει από εκείνο που υπάρχει στο σχέδιο έκθεσης. Το Συμβούλιο συμμερίζεται απόλυτα το στόχο σας να γίνει αυτός ο κανονισμός όσο το δυνατόν πιο φιλικός για τον πολίτη όμως ταυτόχρονα πρέπει να αποτελέσει και ένα αποτελεσματικό και επικοδομητικό εργαλείο. Σύμφωνα με το σχέδιο έξεσης, τα κράτη-μέλη θα κάνουν αυτή τη διαδικασία επιβεβαίωσης των ε, και επικύρωσης των υπογραφών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει στα, στη διάθεσή του τα μέσα επικύρωσης, επιβεβαίωσης των υπογραφών, όλα, όλα δηλαδή την τεχνική υποδομή. Και τον Ιούνιο φέτος κάναμε μακρές συζητήσεις στο Συμβούλιο ε, και είδαμε ότι δεν υπάρχει μία λύση ε, που να ταιριάζει σε όλους. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές νομοθεσίες και τις διαφορετικές δομές σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για την επικύρωση των ε, υπογραφών. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά βάσει των πληροφοριών που έχουμε από τα κράτη-μέλη, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ένα κεντρικό αρχείο του πληθυσμού έχουν κράτη-μέλη άλλα εν συνεχεία διαφορετικά αρχεία και πρέπει να επισημάνουν σε ποια αρχεία πρέπει να ψάξουν για τις κατάλληλες υπογραφές. Ε, σε άλλα κράτη υπάρχουν ε, ταυτότητες, ε, ταυτότητες με συγκεκριμένο αριθμό ταυτότητος. Σε άλλα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν καν ταυτότητες μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ε, δύσκολο για μας να δεχθούμε το παράρτημα 3. Σας επαναλαμβάνω ότι το παράρτημα 3 και η επαλήθευση των υπογραφών είναι δύο πολύ ευαίσθητα ζητήματα και υπάρχουν ε, και άλλοι περιορισμοί στα κράτη-μέλη που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Παραδείγματο χάρη, ελάχιστη ηλικία θέση ε, ενισχύ του κανονισμού αυτού κλπ. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Κομισιόν και τους εισηγητές στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα που θα αποβεί ε, προς όφελος των πολιτών μας. Αυτό επιδιώκουμε άλλωστε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Madame Delcheva is the first one. Είναι η πρώτη συνάδελφος που ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που αφορά την συμμετοχική δημοκρατία. Γιατί και θέλουμε ένα εργαλείο να είναι απλό, να είναι ξεκάθαρο, να είναι προσβάσιμο και να εξυπηρετεί πραγματικά του πολίτε. Να μπορούν να λύσουν τα προβλήματά του. Τώρα, για να δούμε διάφορα θέματα τα οποία ανέκυψαν από τα όσα είπαν Συμβούλη, Επιτροπή και οι εισηγητή. Πρώτα-πρώτα, να σας υπενθυμίσω δύο τεινά τα οποία δεν αναφέρθηκαν. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος εκάλυψε τα όσα είπαμε στην ε, ΛΥΜΠΕ σε σχέση με τη συλλογή υπογραφών όσον αφορά την εθνικότητα και το τρόπο τοποκατοικία, διότι είναι σημαντικό να μπορούν οι Ευρωπαίοι που μένουν σε μια τρίτη χώρα να προσυπογράψουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Όμως, η επιλογή μεταξύ εθνικότητα και τόπου δεν καλύφθηκε από το κείμενο. Τώρα, όσον αφορά τη σχετική προθεσμία, ξέρει ο συγκεκριτής ποια είναι η θέση μου. Είπαμε για αυτό το 12 μήνο. Ναι. Είναι πρώτη σημαντική για τους πολίτες. Να μπορεί κανεί δηλαδή να έχει το χρόνο να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερε ε, υπογραφέ στη δεδομένη ε, προθεσμία. Τώρα άλλα θέματα τα οποία έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά αυτό που μα απάντησε για το εκατομμύριο των υπογραφών των ε, υποβληθισών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανεί να φτάσει εύκολα. Γιατί δεν θα πρέπει κανείς αφού κάποιος υπεγράψει να τους απογοητεύσει και γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει αυτό το τρίμηνο. Άλλωστε έχουμε και το άρθρο 225 της συνθήκης και άρα δεν μπορεί παρά να είναι αυτή η ρύθμιση ικανοποιητική, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικές οι ακροάσεις 14 και 15 που είπαμε ότι θα γίνουν και έτσι θα μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις αυτών που οργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακεί για αυτές τις εκδηλώσεις η Επιτροπή μας. Ήδη έχουμε πάρα πολύ θετικές εμπειρίες, άρα θα πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή με τον κόσμο, οπότε έτσι και εμείς να μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες και να αξιοποιείται ο θεσμός αυτός. Επίσης, σας επισύρω την προσοχή σε άλλα δύο σημεία που είναι πάρα πολύ βασικά όσον αφορά την διαφάνεια για την οικονομική πλαισίωση. Να αποφύγουμε οι πρωτοβουλίες να χρηματοδοτούνται από πολιτικά κόμματα και αν δεν το απαγορεύει ο κανονισμός τότε πολιτικές αρχές που ήδη έχουν ε, μέσα επικοινωνίες και διαφήμισης να μην τους δώσουμε ακόμα ένα όπλο για να προβληθούν. Θα πρέπει με κάθε τίμημα να περιφρουρήσουμε το πνεύμα της ιδέας της πρωτοβουλίας και να είναι έτσι ένα αυθεντικό μέσο συμμετοχής δημοκρατίας. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του κατοφλίου της χρηματοδότησης των πρωτοβουλίων. Δεν θέλω να πω στους ε, συνεισηγητές το εξή. Γιατί να έχουμε αυτό το κατόφλι και κάτω από αυτό θα πρέπει να, να, κάνουμε τη δήλωση του πόθεν έσχες. Το 44 και το 50 αυτές οι διατάξεις αναφέρουν σχετικά. Τι γίνεται με αυτές τις κατεξουδότηση πράξεις και καθορίζεται το κατόφλι. Εγώ πάντως έχω πολλές επιφυλάξεις για αυτές τις διατάξεις. Τι γίνεται κάτω από αυτό το κατόφλι. Υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Εάν έχουμε χίλια ευρώ κατόφλι. Τι είναι αυτό. Είναι από τη μια το ελάχιστο, ελάχιστος μισθός στη Γαλλία, αλλά από την άλλη μεριά είναι τέσσερα μεροκάματα για την Βουλγαρία. Τι γίνεται εδώ. Προσέξτε. Γιατί εδώ είναι θέμα διαφάνειας και θέμα ισότητας μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαίων. Επομένως, έχουμε τόσο που χωρίζουν τους Ευρωπαίους, μην προσθέσουμε ακόμα κάτι άλλο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι πιο αποτελεσματικό το μέσο αυτό. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Ντέλτσεβα. Και τώρα κυρία, κυρία Μπράουν. Thank you very much. I'd also like to... Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για το έργο τους. Νομίζω ότι βασικά βελτιώνει αυτή η προσπάθεια την υποβληθής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση, κυρίως όσον αφορά το ότι εξασφαλίζει ότι το, η εξέταση κατά πόσο ένα αίτημα είναι παραδεκτό γίνεται λιγότερο γραφειοκρατικό, είναι καλή προσέγγιση που προτείνεται. Εγώ υποστηρίζω ένθερμα την πρότασή τους. Είναι σαφές ότι είναι δικαίωμα πρωτοβουλίας παρόμοιο με αυτό που έχει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μ' αρέσει η προτινόμενη διατύπωση στην τελική σκέψη 17 και ελπίζω επ' αυτής της βάσης να προχωρήσουν. Χρειάζεται μεγάλη διαφάνεια, χρειάζεται άνοιγμα, πρέπει να είναι εύχριστο το μέσο αυτό. Και είναι καλό το ότι είναι σαφές το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα το πρωί και θέλω να ακούσω περισσότερα. Θέλω να ξέρω τι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διοργάνωση της ακροάσεως. Είναι σημαντικότατο όμως αν καταφέρουν οι πολίτες να συλλέξουν ένα εκατομμύριο υπογραφές να πάρουν κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο από ότι μια ευχαριστήρια επιστολή στο τέλος. Όσον αφορά σημεία στα οποία αποκλίνω είναι το χρονικό όριο, 24 μήνες θα ήθελα αντί 18. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί, χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Όσον αφορά τον αριθμό των 100 μελών, ίσως είναι καλύτερο να έχουμε αριθμό αντί ποσοστού. Θεωρώ ότι 3 με 4 κάτι μέλη αρκεί. Αυτό θα υποστηρίζαμε ευπρόσδεκτο ότι έγινε κάποια μετακίνηση επί των δύο σημείων, αλλά εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε περισσότερο. Ευπρόσδεκτο το ότι μειώνεται και το όριο ηλικία. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν απαράδεκτη σχετικά με αυτό και εγώ θα προχωρούσα πιο πέρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο ηλικία και θα το υποστηρίξω αυτό. Αν θέλουμε οι νέοι να συμμετέχουν, είναι πολύ σημαντικό να μην θέσουμε όριο ηλικίας πιο λογικό το έντυπο και ο τρόπος συλλογής των υπογραφών. Βέβαια υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ κρατών μελών, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει η υπηκότητα να αναφέρεται στο έντυπο. Εκεί που διαφωνώ περισσότερο και ότι πιστεύω ότι χρειάζεται πιο στεναρή διατύπωση είναι το θέμα της διαμονής. Να εξαιρείται Όταν μιλάμε για την Ευρώπη θέλουμε να είναι κοντά στους πολίτες, εννοούμε μόνο εκείνους που έχουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Ε, στη χώρα μου ε, θεωρούμε ότι είμαστε κοντά στον πολίτη. Στη ΣΥΠΑ λέμε ότι πρέπει να είμαστε κοντά στις βάσεις. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές διατυπώσεις. Θέλαμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Αυτό είναι το νόημα αυτό. τώρα εκείνοι που έχουν άδεια διαμονής και μακράς διαρκείας και εκείνοι που μπορούν να είναι υποψήφοι για δημοτική σύμβουλη δεν μπορούν να υπογράψουν την πρωτοβουλία των πολιτών. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένα φρικτό μήνυμα. Και θα πρέπει αυτό να το θέσουμε στις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεμπρούν. Ο κ. Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια προς τους εισηγητές, εντυπωσιακό το έργο που επετέλεσαν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να είναι παράδειγμα αυτό. Να δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε και στο μέλλον σε παρόμοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, Επί τριών σημείων χρειάζεται, χρειάζονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκή Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, αριθμός κρατών μελών. Δεύτερον, Ποιο έχει το δικαίωμα υπογραφή τη Πρωτοβουλία των πολιτών, διότι όπως μας είπαν στο Συμβούλιο αποκλίνουν οι απόψεις και τρίτον ηλικία και εδώ Καλά το θέτει το Κοινοβούλιο. Καλή είναι η βάση που έχει το Κοινοβούλιο διαπραγματεύσεων του άλλου δύο φορεί για τι ακροάσει. Δεκεκριμένοι συνάδελφοι, πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διστάζει στο να θέσει περαιτέρω διοικητικό άχθος και όχι μόνο επί των νόμων της. Είναι σε καλύτερη θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διοργανώσει την ακρόαση. για έναν προφανή λόγο κατά κάποιο τρόπο εμείς εκφράζουμε την ποικιλομορφία των απόψεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως πολιτικές ομάδες και ως άμεσα αιρετή εκπρόσωποι του λαού. Είμαστε σε θέση να παίξουμε αυτό τον ρόλο. Έχοντας υπόψη και την άποψη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύτοβιτς, εγώ ενθαρρύνω την ιδέα αυτή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το διοργανώνει αυτό. Και θα πρέπει η Επιτροπή Αναφορών εντό αυτού να έχει ένα σαφή διακεκριμένο ρόλο και φωνή. Απευθύνω έκκληση του διακεκριμένου συναδέλφου. Παρακαλώ να αυξήσετε το ρόλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών. Στο τέλος, ένα απλό σχόλιο. Εντάξει, η πρωτοβουλία των πολιτών αφορά την συμμετοχική δημοκρατία. Όμως, φίλοι, συνάδελφοι, αν η συμμετοχική δημοκρατία δεν επηρεάζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές, δεν αλλάζει προς το καλύτερο τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς, αυτό αυτομάτως θα σκοτώσει τις ελπίδες και τα όνειρα των Ευρωπαίων πολιτών μας. Για μένα το σημαντικότερο είναι να επηρεάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές μέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών. Όχι να προσθέσουμε άλλο ένα μέσο, άλλο ένα εργαλείο και στο τέλος να πούμε σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην Ευρώπη «Συγγνώμη, κάτι κάνατε και λοιπόν πρέπει κατόπιν αιτήματό τους να μπορούμε να επηρεάζουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανονισμούς. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Και εξυπηρετώντα αυτό το σκοπό, εξυπηρετούμε και τους Ευρωπαίους πολίτες και τι ανάγκε τους. Και θα συμμετέχουν περισσότερο στις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων οι Ευρωπαίοι πολίτες έτσι. Και ξανά συγχαρητήρια στους διακεκριμένους συνεισηγητές μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποστινάρου. Η κυρία Γκουνιέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μποστινάρου. Θέλω να επιμείνω επί της εμπειρίας Επιτροπής Αναφορών και τη συνάντησή μας με τους Ευρωπαίους πολίτες η Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι μια υπέροχη ιδέα, υπέροχη δυνατότητα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω επί του ρόλου της Επιτροπής Αναφορών και θέλω να ξέρω τι λένε οι συγγητές από αυτού, κυρίω όσον αφορά τη δικασία των ακροάσεων και για την, λάβουμε υπόψη και την εμπειρία που έχουμε όσον αφορά τον απόδεκτο των τιμάτων και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών έχουμε προβλήματα. Όταν καταφθάνει η αναφορά και λέμε στους αναφέροντες δεν είμαστε εμεί αρμόδιοι όσον αφορά την αναφορά σας, βλέπουμε πώς απογοητεύονται. Δεν θέλουμε η πρωτοβουλία των πολιτών να οδηγήσει σε πολλέ απογοητεύσει. Και τέλος όσον αφορά τις πρωτοβουλίες των πολιτών που δεν θα γίνονται αποδεκτές διότι δεν έχουν συλλεγεί αρκετές υπογραφές ή δεν θα εμπίπτουν στα σωστά νομοθετικά πλαίσια. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο ε, το ενδεχόμενο τι γίνεται εκεί και μήπως ε, μπορούμε να βρούμε τη σωστή προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρινή. Και τώρα ο τελευταίο συνεδρός που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε και τους εισηγητές που έβαλαν ένα τόσο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δύο απογοητεύσεις σημειώνονται. Η πρώτη συμβαίνει όταν καθυστερήσει η πρωτοβουλία των πολιτών, διότι υπάρχουν υπογραφές, αλλά αργούν να την υποβάλουν και είναι εκτός προθεσμιών. Ε, οπότε απογοητεύονται πολύ βεβαίως. Και εν συνεχεία, άμα δεν θεωρηθεί αποδεκτή. Θα ήθελα λοιπόν τα κριτήρια να μην είναι υπερβολικά χαμηλά. Έτσι ώστε να έχουμε μία χιονοστιβάδα καινούριων πρωτοβουλειών. Εγώ είμαι υπέρ της ιδέας, υπέρ της ταξινόμησης των πρωτοβουλειών, αλλά όχι να, να μην θέσουμε ένα κατόφλι υπερβολικά χαμηλά, έτσι ώστε όλες οι πρωτοβουλίες να είναι αποδεκτές. Πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε ελάχιστα κριτήρια. Το ελάχιστο που πρέπει να ικανοποιήσουμε τους πολίτες μας είναι να πιστεύουν ότι ακούγονται, ότι ακούγεται η φωνή, η τους. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει η δημόσια ακρόαση δεδομένου ότι η δημόσια φωνή όλων των πολιτών είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν στη δημόσια αυτή ακρόση το σώμα μας πρέπει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι όλων των πολιτών και θα πρέπει να το δώσουμε αυτό στους πολίτες μας να το καταλάβουν, να το δείξουμε. Η άλλη ερώτηση είναι τι γίνεται με, τους, ε, με τις πρωτοβουλίες που είναι τσίμα-τσίμα στο ένα εκατομμύριο δεν είναι αποδεκτές αλλά δεν είναι και τόσο ε, καταρριπτές. Εγώ θα έλεγα να υπάρχει ένα περιθώριο επίκαιας ε, αν δεν μαζευτούν ακριβώς ένα εκατομμύριο αλλά λίγο λιγότερο από το όριο να μπορούμε να τις ε, υποβάλουν στην Επιτροπή Αναφορών. Ο Πρόεδρος. Ωραία, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση θα δώσω το λόγο και στην κυρία Βόλης, αλλά σύντομα παρακαλώ γιατί έχουμε αργήσει. Έχουμε πολλές αναφορές να εξετάσουμε. Ο... Α, κυρία Βόλης πρώτα. Θα είμαι σύντομη. Σα ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια, διότι γενικά ε, κατάλαβα ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Πολλοί συνάδελφοι έσυξαν το θέμα της διαμονής έναντι της υπηκότητας, το θέμα του ορίου ηλικία. Όλα αυτά είναι θέματα και παρακαλώ τους συναδέλφους αν έχουν έντονες απόψεις επ' αυτών να υποβάλω τροπολογίες μέσω των πολιτικών ομάδων διότι πραγματικά εάν έχουν έντονες πεπιθήσεις, χρειαζόμαστε τις τροπολογίες για να έχουμε ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μας στη διαπραγμάτευση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που συνάδελφοι υποστήριξαν τη δική μας επιθυμία να παίξει έναν ηγετικό, έναν δυναμικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα απλώς να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα ζήτημα, όπου πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ε, σωστό ότι η Επιτροπή αυτή πρέπει να παίξει το ρόλο της όταν υπάρχει μια σωστή πρωτοβουλία. Ας προσέξουμε όμως τι ρόλο θέλετε να παίξουμε ή δεν πρέπει να παίξουμε όταν είναι ανεπιτυχής οι πρωτοβουλίες αυτές, όταν δεν περάσουν. Σε αυτές που περνάνε βεβαίως θα παίξουμε το ρόλο μας, αλλά σε αυτές που δεν, που δεν περνάνε, αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν περάσει όλα τα τεστ και θα έχουν κρυθεί ότι δεν είναι κατάλληλες, δεν είναι αποδεκτές. Αυτό που δεν θα ήθελα καθόλου να γίνει σε αυτή την Επιτροπή είναι να γίνει ένα σκουπιδοντενεκές όπου μέσα θα πέσουν όλες οι απο, αποτυχημένες πρωτοβουλίες, οι μη αποδεκτές και μετά θα πρέπει εμείς να τις εξετάσουμε. Δεν λέω ότι οι πολίτες μας έχουν πάρα πολλές επισημίες, πάρα πολλές καλές ιδέες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πρωτοβουλειών που θα κρυθούν αποδεκτές και αυτό που θα κριθούν μη αποδεκτές. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο, μία γραμμή διαχωριστική. Ορισμένα με, μέλη μου είπαν, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, τι θα γίνει, Νταϊάν, όταν ε, αφήσουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες να περάσουν, ε, τι ε, οικονομικό βάρος θα δημιουργήσουμε. Δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία, είναι κάτι καινούργιο που θα γίνει. Αλλά μην ξεχνάτε και το κόστος, έτσι. Ωραία. Αυτά είχα να πω, δεν θέλω τίποτα να προσθέσω, εκτός ε, του να σας ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξή σας, τη συνεργασία σας ε, και τις μελλοντικές μας εργασίες. Ευχαριστώ. No, I Θέλει να συνεχίσει να προσθέσει τίποτα. Όχι, εντάξει, έχουμε ξεκινήσει επισήμως πλέον τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ όλες τις παρατηρήσεις και τις ιδέε ιδέες, τα σχόλια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση μεταξύ του να κάνουμε υποχρεωτικές ακροάσεις από την Κομισιόν αλλά και να διοργανώσουμε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Είναι υποχρεωτικά αυτά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ως Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε να μην μείνει απ' έξω η Κομισιόν. Στην Κομισιόν απευθύνονται, είναι ο βασικός φορέας στον οποίο απευθύνονται οι πολίτες, όμως πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής μας. Αναφορώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα για να πληρώσουμε να σας πενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε 9 η ώρα το πρωί στις 22 Νοεμβρίου 22 Νοεμβρίου στο Στασβούργο για τις τροπολογίες. Α, τροποθεσμία τριπολογιών 15 Νοεμβρίου 6 ώρα. 6 μετά μεσημβρία. Ωραία, προχωρούμε λοιπόν. Είναι η ε, αίτηση... υπάρχουν 7. Την έχει υποβάλει ο Βάλτερ Γκρίτσικ. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Έλεγα ότι έχουμε την αναφορά επαριθμών 7 του Βάλτερ Γκρίτσικ. Ε, είναι ε, ένα πρόσωπο γερμανική ηθαγένεια για λογαριασμό του Γκίντερ Μόντελγεν σχετικά με την παραβίαση τη οδηγία 2003 κάθετο 8 του Συμβουλίου για το ευεργέτημα τη παινία σε διασυνοριακέ διαφορέ. Παρίσταται ο αναφέρον. Όχι, τότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Βικτορόβιτς, πώς λέγεστε, δεν ξέρω αν λέω καλά το όνομά σας. Thank you very much. Uh, petition... Εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτή η αναφορά αφορά κάποιο πρόβλημα. πράγμα τη ιδιοκτησία στην Ισπανία έχουμε κάποιον ο οποίο ζήτησε το ευαγγέλιο τη παινία να καλυφθούν τα οδηπορικά του όσον αφορά την ε, εκδίκαση διαδικασία σε δικαστήριο Ισπανικό. Καταρχήν ε, ίσως ε, αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση με την οδηγία αυτή του 2003 κάθετος 8, ιδίως δυνάμει του άρθρου 7. Όμως ε, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ορθό, διότι αυτή η οδηγία μόνο ορίζει ε, ποιες δαπάνες θα καλύπτονται σε σχέση με τη χορήγηση του ευεργετήματος παινίας και δεν ισχύει όσον αφορά κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν χορηγεί το ευεργέτημα παινία. Οπότε πρόκειται για ρύθμιση που γίνεται από το εθνικό δίκαιο και σε συγκεκριμένη περίπτωση από το ισπανικό δίκαιο, όπως ορίζουν τα άρθρα 12 και άρθρο 5. Και για αυτού του λόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας προτείνει να κλείσει η αναφορά. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Wanted the floor about this issue. Θέλετε το λόγο. Α, είναι εδώ αναφέρον και νόμιζα ότι δεν ήσασταν εδώ. Ο κύριος Γκρίτσι Μίλησε η Κομισιόν, αλλά θέλετε εσείς το λόγο. Ναι, σας, σας είπα. Ε, έπρεπε να βγω για δέκα λεπτά. Επισημούσα έτσι λίγο πιο μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί μόνο μία αναφορά μπόρεσα να προβάλλω Λοιπόν, το ερώτημά μου θα ήταν κατά πόσον όταν δίνουμε ενίσχυση οικονομική για την περαίωση των διαδικασιών, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία διαδικασία. Δεν έχω την εντύπωση ότι ε, ε, επειδή υπάρχουν διαφορετικές, ε, ε, διαφορετική διαμόρφωση των τιμολογίων, παραδείγματο χάρη τιμολόγια από δικηγόρους, τιμολόγια από άλλους φορούς, έχουμε μία ικανοποιητική διαχείριση όλων αυτών των διαφορετικών τιμολογίων και λογαριασμών. Και διαφέρει, ας πούμε, και το κόστος υπηρεσιών σε μια χώρα σε μια χώρα είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος υπηρεσιών, σε άλλες χώρες είναι, είναι χαμηλότερο το κόστος. Οπότε, ε, παραδείγματο χάρη, όταν κρίνω εγώ το εισόδημα ενός ε, ετούντος, ε, καταλήγω σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα από ότι ε, ένας άλλος υπήκος, ένα άλλο κράτος μέλος, ο οποίος θα είχε ένα διαφορετικό εισόδημα, διαφορετικό μισθό. Έχουμε λοιπόν και τα μισθολόγια και το κόστος σε πολύ διαφορετικό επίπεδο. Τι θα γίνει λοιπόν με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης τους ετούντες αυτούς που δεν έχουν τα μέσα να προχωρήσουν τη διαδικασία με κόστος από την τσέπη τους. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τι, τα διαφορετικά επίπεδα ε, κόστους ε, τιμαρίσμου στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη, στο Λουξεμβούργο καμία διαδικασία δεν θα λάμβανε οικονομική ενίσχυση γιατί το βιωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, ενώ και όταν, αν ένα υπήκοο από το Λουξεμβούργο έχει μια ε, δικαστική διαδικασία σε ένα άλλο κράτο μέλο με χαμηλό κόστο ζωή, δεν θα τον ενισχύαμε ποτέ, διότι θα προερχόταν από μια χώρα με υψηλό εισόδημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαμορφωθούν και βάσει της ισπανικής παρέμβασης διάφορες συντελεστές εξομάλυνσης των διαφορών αυτών για να μην υπάρχουν αδικίες σε ποιους παρέχουμε αυτή τη νομική βοήθεια. Ευχαριστούμε κύριε Βιλάν. Ναι, δεν προβλεπόταν να μιλήσετε, αλλά έτσι όπως ετέθη το θέμα τώρα πρέπει να σας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε και κάτι να πείτε κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η οδηγία ρυθμίζει μόνο συγκεκριμένη διαδικασία. Και περιορίζεται στο να ορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ευεργέτημα παινίας χορηγείται. και βέβαια χορηγείται από εθνικές αρχές, εθνικά δικαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ή στη συγκεκριμένη χώρα. Γιατί αυτό αφορά το ευεργέτημα παινίας και καλύπτονται οι περισσότερες από τις δικαστικές δαπάνες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ισότητα μεταχείρισης για όλους τους Ευρωπαίους. Mr. habe ich das richtig verstanden? Συγγνώμη, σας κατάλαβα καλά ότι η οδηγία εγγυάται ότι κάποιος που ότι κάποιος ο οποίος περνάει από μια διαδικασία δικαστική σε μια άλλη χώρα δικαιούται, καλύπτεται από τη βοήθεια αυτή, από την ε, ενίσχυση αυτή. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω είναι ότι ίσω θα πρέπει να σα παραθέσω το άρθρο 5 παραγωγή 3 τη οδηγία, διότι εκεί άμεσα σα καλύπτει σε αυτό που είπατε. Εκεί ορίζεται τα κράτη-μέλη. Είναι δυνατόν να ορίζουν κάποια κατόφλια κάτω από τα οποία ε, θεωρείται ότι κάποιο δικαιούται ε, το, το, το, το ευεργέτημα παινία. Αυτό ορίζει. Επιλέξει η οδηγία. Οπότε και εγώ δεν έχω τίποτα να σας πω γι' αυτό. Bien, señor Κύριε Βιλάν, θέλετε να δευτερολογήσετε. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε κι άλλο. Δεν είμαι ικανοποιημένο. Το ότι υπάρχουν ε, συγκεκριμένα κατόφλια παρέμβαση σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν, το ξέρω. Εάν σε ένα κράτος μέλος έχει μέσο εισόδημα 2.000 ευρώ, και ένα άλλο κράτος μέλος όπου γίνεται η εκδίκαση, το μέσο, ο μέσος ε, όρος μισθού είναι 1000 ευρώ, κάποιος ξεκινάει μια δικαστική προσφυγή που προέρχεται από ένα άλλο κράτος μέλος όπου ας πούμε ο υπήκοος που κάνει την ε, προσφυγή, τη μήνυση έχει, προέρχεται από ένα κράτος με 3.000 ευρώ μέσο μισθό και ξεκινάει τη διαδικασία σε ένα κράτος με χίλια ευρώ μέσω, μέσω μισθό. Ε, ε, εάν δούμε λοιπόν τη διαφορά αυτή ε, κανονικά στη χώρα προέλευσής του θα ε, δεν θα ελάμβανε ενίσχυση αλλά στη χώρα ε, της προσφυγής θα λάμβανε ενίσχυση ή αντίστροφα αν προέρχεται από πλούσιο κράτος δεν δικαιούται αν προέρχεται από φτωχό κράτος δικαιούται ακόμα και αν το κράτος προσφυγής είναι πλούσιο τι ισχύει λοιπόν, λαμβάνουμε υπόψη το μέσο όρο κόστου ζωής και εισοδήματος στη χώρα προέλευσης ή στη χώρα προσφυγής και εκδίκασης. Ή τρίτη εναλλακτική λύση είναι ότι αναγνωρίζουμε τη διαφορά στη διαβίωση και στο κόστος ζωής και γι' αυτό χρησιμοποιούμε έναν συγκεκριμένο δίκτυ εξομάλυνσης. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν, είναι πρόθυμη να εξετάσει αυτό τον τρίτο δρόμο ε, και να εκδώσει μία καινοτομική ε, απόφαση, μια καινούρια ιδέα, ένας καινούριος δρόμος. Οπότε θα έπρεπε ο ετών να λάβει ενίσχυση παινία στην Ισπανία. Ή πιστεύει η Κομισιόν ότι οι διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη-μέλη είναι δίκαιες και δεν δημιουργούνται ανισότητες και αδικίες μεταχείρισης των πολιτών. Κοιτάξτε, πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, σας υπενθυμίζω αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Είναι σαφές το θέμα. Προτίθεστε ή όχι να μεταβληθεί το αίτημά σας ιδάλλως, θα κλείσουμε την αναφορά. Σε αντίθετη περίπτωση θα περιμένουμε από τη Επιτροπή κρατώντα την αναφορά ανοιχτή, λέει ο Πρόεδρο. Θα ήθελα να απαντήσω πολύ σύντομα σε αυτό. Η οδηγία. Κλείνει το μικρόφωνο του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μικρόφωνο του Κριστο. Η οδηγία στο άθρο 5,4 προβλέπει την περίσταση που μόλις περιγράφει. Οπότε ο αναφέρον μπορεί να προσπαθήσει να αποδείξει ότι τα μέσα που διαθέτει μάλλον ότι μπορεί να δεχτεί νομική ε, αρρωγή παρόλο που δεν ε, είναι εντός του Αλλά το Εθνικό Δικαστήριο θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση. Και αυτή η αξιολόγηση δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της ε, οδηγίας. Άρα λοιπόν θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτό ο φάκελο τη αναφορά και η Κομισιόν να μα πει, εάν, ε, να μας απαντήσει δηλαδή, εάν είναι πρόθυμη να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία ρύθμισης αυτής της ε, παρατυπίας. Ωραία, αυτό είναι δικαίωμά σα, αν το ζητήσετε. Όμω, σα ξεκαθαρίζω ότι θα μην ανοιχτή η αναφορά και άρα θα ζητηθεί και θα αναμένεται πάνω σε αυτό που είπατε η απάντηση της Κομισιόν. Κυρία Γουόλης, έχετε το λόγο. Πολύ γρήγορα να πω ότι κατανοώ τον στόχο του κ. Βίλαντ και συμφωνώ με αυτόν. Ίσως να πρέπει να συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και πολιτικών ελευθεριών. Να διαπιστώσουμε ακριβώς ε, πώς λειτουργεί, πώς εφαρμόζεται, τι καλύπτει αυτή η οδηγία. Εάν συμφωνείτε, σύμφωνα με την πρόταση Wallis, θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να διαβιβάσει το αίτημα στην Επιτροπή, να μελετηθεί το αίτημα και να ληφθεί η σχετική απόφαση. Συμφωνείτε, συνάδελφε. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Έχει να κάνει με τις εξωτερικές σχέσεις. Έχουμε τρία σημεία, τρεις αναφορές, διορθώνει ο Πρόεδρος. Να τα δούμε από κοινού. Είναι τα σημεία 8 και 9. Δύο και όχι τρία όπως λέει ο Πρόεδρος. Ξεκινάμε από το 9 και όχι από το 8. David Peck, Βρετανική Σταγένεια York, εκστρατεία αλληλεγγύη τη Παλαιστίνη και την ανανέωση τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ισραηλινή Επιτροπή κατά τη κατεδάφιση σπιτιών. Και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο David Πέγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή για τη δυνατότητα που μου δίνει για να αναφερθώ στο θέμα του ICAT για μια ακόμη φορά. Αν δεν ξέρετε τι είναι ICAT, είναι η Ισραηλινή Επιτροπή κατά της ε, κατεδάφισης σπιτιών, δημιουργήθηκε το 1997, είναι μια απάντηση μη βία, άμεσης δράσης όσον αφορά την ε, καταστροφή ε, Παλαιστινιακών κατοικιών στην κατεχόν Παλαιστινιακή περιοχή από τους Ισραηλινούς. Από το 1967 τουλάχιστον 24.813 σπίτια καταστράφησαν και δεκάδες χιλιάδες αντιμετωπίζουν την προοπτική της καταδάφισης. Η ICAT έχει ανοικοδομήσει περίπου 170 από τα σπίτια που ίσως να θεωρείται ότι είναι σταγόνα το ωκεανό και από πλευρά ανθρωπιστική είναι κάτι τέτοιο, εκτό για τι οικογένειε, βέβαια, αλλά αντιπροσωπεύει 170 πράξει κοινή αντίσταση από Ισραηλινούς και Παλαιστινίου που συνεργάζονται και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικότατο. Η ανοικοδόμηση σπιτιών, σπιτιών οικονομικών είναι, έχει μεγάλη συμβολική συνέπεια και αξία και η ψυχολογική και θέλει ΆΙΚΑΤ να ενθαρρύνει ενεργό συμμετοχή Ισραηλινών, Παλαιστινίων και κοινωνίε των πολιτών αυτών και τη διεθνού κοινωνίες των πολιτών και να δημιουργηθούν νέε δυνατότητε για μια δίκαιη ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε προγράμματα ICAT το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι το 2007 και το Φεβράριο του 2008 η ΆΙΚΑΤ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος Συνεταίρη για την Ειρήνη συνεργασία την ειρήνη για να αυξήσει τις δραστηριότητε βοήθειας και παιδείας και τις δυνατότητες ανοικοδόμησης. Τον Ιούλιο του 2008 αυτή η αίτηση που είχε υποβληθεί απερίφθη και η συνοδευτική επιστολή με την απόρριψη ανέφερε ότι η αίτηση πληρούσε τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια που απαιτούνται για μια θετική απόφαση και η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε δώσει 80 με 95% μέχρι πλήρη βαθμολόγηση για όσε πτυχέ εκτό από ένα σημείο που αφορούσε τη μεθοδολογία και αφιερωνόταν στην θεωρούμενη ε, μη συμμετοχή επαρκή των Παλαιστινίων εταίρων. Μετά από την ακρόαση που έλαβε χώρα ε, το Σεπτέμβριο, ήρθαμε σε επαφή με τον Μάικλ Ντόχερτη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγιναν πολύ επικοδομητικές ε, συζητήσεις μαζί του και ήταν σαφέστατο ότι παρόλο που η ICAD επί σειρά ετών και με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω εργάστηκε αποτελεσματικά, χρησιμοποιούσαν επίσημε επαφέ με πολλέ Παλαιστινιακέ οργανώσει, η ICAD έπρεπε να εξασφαλίσει πιο επίσημε διασυνέσει με αναγνωρισμένου οργανισμού Παλαιστινιακού, ώστε να μπορεί να πληρεί τι προποθέσει του Partner for Peace. Αυτό έγινε και μια κοινή αίτηση με μια οργάνωση που ήδη είναι καταχωρημένη στο Παλαιστινιακό Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβληθεί στο, στο πρόγραμμα Partners for Peace πολύ σύντομα. Και πρέπει να πω ότι η βοήθεια του Μάικλ Ντόχερ της διοργάνωση όλων αυτών είναι κάτι που εκτιμούμε πολύ. Αυτή η επαφή με τον Μάικλ μας έδωσε τη δυνατότητα επίσης να αποστηρίξουμε άλλη μια πρόταση του ICAT στα πλαίσια του IDHR και της σχετικής πρωτοβουλίας και η χρηματοδότηση διατέθη μετά από αυτή την αίτηση για το πρόγραμμα. Και υπάρχει άλλη μια πτυχή της χρηματοδότησης του ICAT που θα ήθελα να τονίσω. Εν συντομία, είμαι επιστήμον ερευνητή που βασίστηκε στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για το μεγαλύτερο τμήμα τη δουλειά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο και Μία αποτελεσματικό είναι να κινείται κανεί μόνο και μόνο με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Δηλαδή, να, χωρίς να υπάρχει συγχρηματοδότηση. Δηλαδή, χρηματοδότηση η οποία να καλύπτει τι συνεχεί βασικέ υποδομέ για τη δραστηριότητα που απαιτείται. Η ICAD ε, χρειάζεται κάτι παρόμοιο και όπω αναφέρεται στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λέει ότι ε, επαναλαμβάνω το θεσμό μα για το έργο που τελεί η ICAT η συγχρηματοδότηση δεν θα έπρεπε να αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να την υποστηρίζει και να μην τελικά μειώνει την ταχύτητα εφαρμογή του προγράμματο κάθε φορά υπάρχει κενό χρηματοδοτήσεω. Και τέλο, θα θέλαμε να κάνουμε το εξή σχόλιο, απευθυνόμενο στην Επιτροπή. Είναι πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να υποστηρίζει την λύση δύο κρατών όσον αφορά το πρόβλημα Παλαιστινίων Ισραηλινών, αλλά αυτό εμποδίζεται από τι δράσει των Ισραηλινών επιτόπου και κυρίω από την καταστροφή ιδιοκτησία Παλαιστινίων και υπηρεσιών των Παλαιστινίων και την κατάκτηση κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών. 16 χρόνια ε, έχουν δείξει ότι μόνο διαμαρτυρίε δεν ε, λειτουργούν όσον αφορά το Ισραήλ και ήρθε η όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα και ένα κομμάτι αυτό θα μπορούσε να κάνει θα ήταν ένα παροχή σταθερής χρηματοδότησης για το έργο της ICAD. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα δώσω το λόγο το λόγο συγγνώμη στον κύριο Μάικλ Ντόχερτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια της ICAD. Δεν υπάρχουν πολλά να προσθέσουμε σε αυτά που είπαμε πέρσι και αυτά που είπε ο καθηγητής Πέγκ ε, τώρα. Νομίζω ότι καταφέραμε να δείξουμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν χρηματοδοτήθηκε ο ΆΙΚΑ το 2007 δεν οφειλόταν στην ε, επιρροή άλλης ζωηνής οργανώσεως που είχε υποβάλει μήνωση ε, κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει τη οδηγία 1004. Το Σεπτέμβριο είχαμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή Αναφορών πέρσι αυτό το θέμα και καταφέραμε να δώσουμε συμπροματικό ποσό στην αντιπροσωπεία στο Ισραήλ για το IDHR, ε, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε άλλα δύο προγράμματα, ένα από τα οποία ανήκε στην ICAT. Οπότε είμαστε άλλοι αρκετά ικανοποιημένοι, παρόλο που δεν είναι το ίδιο πρόγραμμα όπως αυτό που είχε προταθεί το 2007 αυτό το πρόγραμμα που αφορά τις κατεδαφίσεις των σπιτιών θέλει να σταματήσει αυτές τις κατεδαφίσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα κατεχόμενα εδάφη που εφαρμόζονται σπινές αυτές τις κατεδαφίσεις σπιτιών. Στη Ραμάλα συνάντησα την κυρία Φάντουα Αλσάρ, που είναι επικεφαλή του Υπηρεσία Καταγραφή Μη Κοινωνιστικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών τη Παλαιστίνη και θέσαμε το θέμα τη μη καταχωρήσεω του εταίρου του ICAT, προτιμά ο ICAT, και άλλα θέματα που είχαμε. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν λάβαμε απάντηση, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε κάποια απάντηση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα παρά να το θέσουμε το θέμα. Αυτό είναι ε, θέμα εσωτερικό για την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά το θέσαμε το ζήτημα ότι υπάρχουν μακρές καθυστερήσεις όσον αφορά την καταχώρηση αρκετών ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τον επόμενο χρόνο, από το 2011 μέχρι το 2013, ε, καταφέραμε να πετύχουμε αύξηση χρηματοδοτήσεω τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία του Ισραήλ από 900.000 στα 1,2 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε ελπίζουμε ότι αυτό θα χρηματοδοτήσει ένα-δύο προγράμματα παραπάνω, ένα-δύο τις παραπάνω. Ένα πρόβλημα που έχουμε βλέπετε είναι ότι από τη μία είναι καλό βέβαια το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι όποτε έχουμε αιτήματα, αιτήσει από μη κυβερνητικέ οργανώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, έχουμε πολλέ αιτήσει από εκεί. Και το φράγμα πρέπει να υπερπηδήσουμε. Το εμπόδιο εκεί είναι πολύ πιο ψηλό από τι άλλε χώρε. Λοιπόν, για τη χρηματοδότηση την ε, βασική την, ε, ε, είναι κάτι που υποστηρίζω. Ταιριάζει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση διμερούς συνεργασίας. Χρειαζόμαστε υποστήριξη οικονομική, αλλά θα πρέπει η αρχή του προπολογισμού ασχοληθεί με το θέμα, διότι παραπέμπουμε στη νομική βάση των δράσεων και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος, η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την απάντησή της. Γιατί πολλοί από εμά θα έλεγα σοκαριστήκαμε όταν ακούσαμε ότι αυτή η Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση έχει επιρροή. Ήταν λοιπόν για μας σοκ να δούμε ότι μία οργάνωση όπως η ICAT ήταν απούσα. Πολλοί από μας κατά τη διάρκεια των ετών ε, ε, τους συνεργαστήκαμε, τους ξέραμε. Όταν πηγαίνουμε από τη Δανία στην Ιερουσαλήμ, του ε, τους συναντούσαμε. Ήταν λοιπόν ένα σοκ να μάθουμε ότι δεν, δεν ήταν εκεί. Ε, είμαι ευτυχής τώρα που ακούω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί ένα από τα πολλά ζητήματα σε αυτό το θέμα είναι ότι εμείς πληρώνουμε, πληρώνουμε και δίνουμε συνέχεια λεφτά και αυτή συνέχεια καταστρέφουν, καταστρέφουν. Ε, μία πλευρά καταστρέφει, η άλλη πλευρά πληρώνει, εμείς δηλαδή. Όταν καταστρέφουν λοιπόν στα... We should pay, not our, our taxpayers στα κατεχόμενα θα πρέπει ήδη να πληρώσουν την ανακατασκευή, όχι άλλοι. Αλλά όλοι μας ενεργούμε νευρικά, φοβισμένα, ε, μην τυχόν και πονέσουμε το δαχτυλάκι του Ισραήλ, μην τυχόν και πετήσουμε τον κάλο του Ισραήλ, μην τυχόν και σημώσει το Ισραήλ. αφού αυτοί καταστρέφουν, αυτοί να νοικοδομήσουν και όχι να πληρώνουμε εμείς την ύφη συνέχεια. Άρα λοιπόν να περικόψουμε τα χρήματα που δίνουμε. Εγώ υποστηρίζω πλήρως αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση. Για να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω ο κύριος ε, Περ, ο αναφέρον ζητεί το λόγο. Ο κύριος Πέγκ, ο κύριος Πέγκ. Εντάξει. Ε, νομίζω ότι είπα αυτά που έπρεπε να πω. Ευχαριστώ πολύ και την ε, Μάργαρετ για την ε, υποστήριξή της. Μας ενισχύει πραγματικά αυτό το σημείο της συνεχούς χρηματοδότησης πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστεί από την Κομισιόν. Ε, είναι επίγον πραγματικά πρέπει να, να, να, να εμελετήσει τι γίνεται με, αυτό το θέμα. Συνεχώς στέλνουν λεφτά, συνεχώς γκρεμίζονται οι οικισμοί εκεί, κάτι πρέπει να γίνει. Έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα να κλείσουμε την αναφορά, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Πολύ ωραία. Η άλλη αναφορά. Πάλι αφορά τι σχέσει και υποβληθεί από την Αν Χάλαμ, Βρετανική Ιθαγενεία εξ ονόματος της Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign. Συνοδευόμενο πάντα και υπογραφές και με τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ Ισραήλ. Ο κύριος Πούστερμαν ζητεί το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτή την επιτροπή μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την αναφορά εκ μέρους της διοργάνωσης αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη από το Brighton και το Hove. οι πολίτες της Ευρώπης ή ένα μεγάλο μερίδιο της Ευρώπης αρχίζουν πλέον και αγανακτούν με την έλλειψη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους και με την καταπάταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς Ισραήλ για να μπορέσουμε να βρούμε μία δίκαιη λύση, η, λύση, η βοήθεια για που χρειάζεται δεν θα προέλθει από το εσωτερικό των δύο ενδιαφερομένων μερών, αλλά χρειάζεται τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Αλλιώς δεν θα βρεθεί ποτέ λύση και δεν θα σταματήσουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να παρέμβει δραστικά με όλες τις, τις ε, δυνάμεις για να επιβάλλει μία αναστολή, πάγωμα της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το άρθρο 2 της ε, ε, Συμφωνίας Σύνδεσης Ισραήλ-Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης παραβιάζεται συνέχεια η, άποψη των νομικών εμπειρογνωμόνων είναι ότι εάν δεν λάβουμε μέτρα κατά του Ισραήλ και μετά από τις πρόσφατες βιαιότητες που έκανε το Ισραήλ, ε, η συμφωνία αυτή πλέον θα είναι καινού περιεχομένου, καινή περιεχομένου. Βλέπουμε συνέχεια εκτός από την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ παραβιάζει το άρθρο 11 των ε, συνθήκων, στην οποία βασίζεται αυτή η συμφωνία σύνδεσης. Καταπατάει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ελευθερία και η κυβέρνηση του Ισραήλ αγνοεί συνεχώς τα δικαιώματα και τα αιτήματα των Παλαιστινίων και όσον αφορά οικονομικά και πολιτικά ε, ζητήματα. Επίσης, το Ισραήλ έχει καταφέρει να εξαιρείται από όλες τις ε, νομοθεσίες, από όλες τις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες δεν σέβεται. Το άλλο, ο άλλος λόγος υποβολής της αναφοράς ε, είναι το κόστος προς τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Βάσει της εμπορικής συμφωνίας, ε, τα Ισραηλινά προϊόντα επιδοτούνται εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εισάγονται. Ε, πολλά προϊόντα που εισάγονται μέσω Ισραήλ και έτσι απαλλάσσονται εν μέρη από δασμούς βάσει της πλεονεκτικής αυτής συμφωνίας το 2009 500 εκατομμύρια ευρώ η Κομισιό ταξόδεψε στα κατεχόμενα. Δίνουμε πολλά λεφτά, εκατομμύρια ευρώ στα κατεχόμενα, όμως δεν μας καταβάλει το Ισραήλ καμία αποζημίωση για την καταστροφή των έργων αυτών τα οποία εμείς χρηματοδοτούμε στα κατεχόμενα. Δηλαδή, καταστρέφει οικοδομές, σπίτια, οτιδήποτε στα, υποδομ, στα υποδομές, στα κατεχόμενα, τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς, αλλά δεν έχουμε ποτέ πάρει μία δεκάρα αποζημίωσης από το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν διακυβεύεται το καλό όνομα της εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται ότι εμείς επιβραβεύουμε το Ισραήλ για αυτά τα οποία γίνονται στη λωρίδα της ε, Γάζας. Όλες οι διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν αποφέρει μηδαμινό αποτέλεσμα και ο Παλαιστινιακός λαός αισθάνεται εγκαταλελειμμένος και αφημένος στη μοίρα του όλη η πολιτική της επιβολής της ειρήνευσης στην περιοχή αυτή επί 62 χρόνια όχι μόνο έχει αποτύχει πλήρως αλλά βιαιότητες και γενοκτονία συνεχίζεται και μάλιστα έχουν οξυνθεί τα φαινόμενα και καταδικάζονται διεθνώς. Γι' αυτό πρέπει και ζητούμε, κάνουμε μια έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει κάθε προσπάθεια να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική προς το Ισραήλ, να παγώσει η, συμφωνία, η εμπορική συμφωνία Ισραήλ-EU και να τιμωρηθεί το Ισραήλ βάσει του, του διεθνούς νόμου, του διεθνούς δικαίου, συγγνώμη. Κυρία Μπούστρεμαν, σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρικάρντο Σάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Χάλαμ. Είμαστε γνώστες του θέματος και των ε, απόψεων που εκφράσατε. Όχι ότι συμφωνούμε απόλυτα με την ανάλυση σας και δεν συμφωνούμε και με τις ε, ποινές ε, που προτείνετε. Βεβαίως υπάρχει μία ρήτρα στην συμφωνία, στην υπάρχουσα συμφωνία που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως η συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ όπως και με άλλες χώρες στα πλαίσια της ε, πολιτικής ε, καλής γειτονίας μας υποχρεώνουν να έχουμε καλές ε, σχέσεις. Πιστεύω ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ακριβώς δεν πιστεύω ότι το πάγωμα αυτής της συμφωνίας θα είναι ε, ωφέλιμη και για, για, για μας, για τη δική μας πλευρά. Εμείς έχουμε αντίθετη άποψη. Εμείς πιστεύουμε ότι η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελεί τη βάση του διαλόγου, του διαλόγου με το Ισραήλ και αυτός ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί αν θέλουμε να επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε και πολλές εναλλακτικές λύσεις παρά το να εκφράζουμε στο Ισραήλ τις επιφυλάξεις μας, τις αντιρρήσεις μας και όλα αυτά τις απόψεις δικές μας μπορούμε να τις εκφράσουμε μόνο μέσω των τακτικών συνεδριάσεων που ορίζονται από αυτή την εμπορική συμφωνία. Παραδείγματο χάρη, το Σεπτέμβριο είχαμε μία συνεδρίαση τη υποομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συζητήσαμε σε βάθο αυτό το θέμα και το Δεκέμβριο πάλι θα συνεδριάσει αυτή η υποεπιτροπή και στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου μπορούμε να εκφράσουμε εμείς τις αντιρρήσεις μας ή τις παρατηρήσεις μας ε, προς το Ισραήλ ε, χωρίς ε, να και να, γίνουμε, να μας ακούσουν κιόλα. Εάν ε, με αυτή την συμφωνία πλαίσιο την καταργήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το τακτικό διάλογο. Και πώς θα ακούγονται οι απόψεις μας. Καταλαβαίνω το δίλημά σας βεβαίως. Αυτή είναι όμως η θέση μέσα στην οποία βρισκόμαστε και η θέση δικιά μας διαφέρει από τη δική σας. Προσπαθούμε στις σχέσεις μας με το Ισραήλ να εδραιώσουμε ορισμένα κριτήρια μη Ε, Παραδείγματο χάρη, η αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ δεν έχει συμβεί, έχει, έχει παγώσει. Βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο σχέσεων, ενώ υπήρχε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι μπορούμε να αναβασμίσουμε τις σχέσεις μας μόνο αν έχουμε στοιχεία, αν μας αποδείξουν ότι έχουν προχωρήσει στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε ε, βήμα προς βήμα, αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που ισχύει με το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βόλης έχει το λόγο. Κυρία Βόλης, όχι. Ο κύριος Τέιλορ. Πρώτα στην κυρία. Είσαστε κύριος και δίνουμε το λόγο πρωτίστως στην κυρία. Δεν ήθελα να μιλήσω πριν από τον κύριο Τέιλορ, δεν επέμενα, αλλά ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, ήθελα να κάνω μια σειρά παρατηρήσεων μετά από αυτά που άκουσα από την Κομισιόν. Ήμουν ε, ένα από τα μέλη που μελέτησα με προσοχή την νομική γνωμοδότηση ενός Βρετανού νομικού για το αν υπάρχουν λόγοι και επαρκές, ε, επαρκή στοιχεία να προσφύγουμε κατά του Ισραήλ για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω λοιπόν εξετάσει με μεγάλη γνωμοδότηση. Και από ό,τι καταλαβαίνω η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν θέλει να προβεί να προχωρήσει νομικά με, με δικαστικά βήματα ή με προσφυγές. Όμως υπάρχουν πολλά καυτά θέματα και η Κομισιόν μας είπε ότι μελέτησε με μεγάλη προσοχή τη νομική γνωμοδότηση. Η νομική αυτή γνωμοδότηση λέει σαφέστατα ότι όχι μόνο το Ισραήλ έχει υποχρεώσεις να σεβαστεί ορισμένα πράγματα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει όταν βλέπει ότι ένας από τους εταίρους της με τον οποίο έχει μία συμφωνία παραβιάζει τις ε, συνθήκες, παραβιάζει τις διατάξεις της συμφωνίας. Δεν ξέρω τώρα, εάν υπάρχει δυνατότητα ένα συγκεκριμένο σώμα, μία επιτροπή παραδείγματο χάρη, να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτή της νομική γνωμοδότηση, την οποία έχουμε στα χέρια μας. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ μία εξέταση αντικειμενική από μία άλλη επιτροπή. Βεβαίως, τα όσα έχουν γίνει στη λωρίδα της Γάζας είναι προφανή και είναι, οι βιαιότητες αυτές ε, είναι ε, φοβερές. Ε, όμως, οι διοκτήτες και Παλαιστίνοι πολίτες που δεν είναι μόνο στη λωρίδα της Γάζας συνεχώς υποφέρουν επειδή δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα, τους τα δικαιώματά τους. Ο Παλαιστίνοι πολίτες, οι ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν γκρεμιστεί και αλλού λοιπόν συνεχώς θίγονται. Άρα πιστεύω ότι υπάρχουν εκεί πολίτες που μπορούν να αναλάβουν μεμονωμένη δράση και να υποχρεώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει. Οπότε εκεί θα βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ. Θα απαντούσα, στην Κομισιόν λέγοντας, ε, επειδή είπε η Κομισιόν ότι δεν θέλει το πάγωμα της συμφωνίας κλπ. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή τους, δίνει, τους παρέχει ένα εργαλείο διαλόγου. Αυτό είπε η Κομισιόν αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς τώρα παρόντας στην Κομισιόν είναι ότι αυτό το εργαλείο έχει πάψει να λειτουργεί πια. Είναι εκτός λειτουργίας. Αν δείτε πώς συμπεριφέρεται το Ισραήλ σε σχέση με την Παλαιστίνη. Αυτή η αναφορά δεν είναι εναντίον του Ισραήλ, αλλά είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Είναι μια αναφορά που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Και πιστεύω ότι εμείς το Κοινοβούλιο πρέπει να την κάνουμε αποδεκτή. Εάν δεν υπεραμεινόμεθα του διεθνούς δικαίου, ε, τι κάνουμε τότε. Θα ήθελα να παρέμβω και να ε, αναφέρω ένα άλλο γεγονός πριν από δυόμιση χρόνια η κυρία Χάλαμ που προέρχεται από την εκλογική μου περιφέρεια υπέβαλε μια άλλη αναφορά. Ε, μια άλλη αναφορά. Δυόμιση χρόνια βρίσκεται πάλι εδώ, σχεδόν έχουμε 2011 με το ίδιο θέμα. Η Επιτροπή λοιπόν τότε είχε κάνει αποδεκτή την αναφορά και την παρέπεψε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων. Αυτό έγινε τον Ιούλιο 2009. Την παρέπεμψε λοιπόν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, διότι ήταν η πιο κατάλληλη επιτροπή να απαντήσει. Όμως, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν έχει, ε, υποθέσεων, δεν έχει μελετήσει καν την αναφορά, το ζήτημα. Άρα λοιπόν, από τον Ιούλιο του 2009 η αναφορά αυτή των πολιτών του Brighton και Hove εκρεμεί. Καταλαβαίνω ότι το θέμα αυτό διχάζει Καταλαβαίνω ότι όποτε συζητιέται η συζήτηση είναι δύσκολη, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε κολλήσει. Είμαστε σε ένα αδιέξοδο, έχουμε κολλήσει, δεν έχει προχωρήσει τίποτα με αυτή την αναφορά. Άρα λοιπόν το ερώτημα τίθεται, τι πρέπει να κάνει αυτή η Επιτροπή Αναφορών. Κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση αυτή του αδιέξοδου ηρωνεύεται τη λειτουργία μας, μα, μας κοροϊδεύει, ε, λέει, μας λέει κατάμουτρα, μα τι κάνετε εσείς εδώ αφού δεν μπορείτε να προχωρήσετε αυτό το, αυτή την αναφορά. Ε, δεν λέω ότι θα πρέπει να δώσουμε ε, ουτοπικές προσδοκίες τους ετούντες, αλλά εν πάση περιπτώσει μια αναφορά που έχει κολλήσει δύο χρόνια σχεδόν και δεν προχωράει, είναι μια κοροϊδία τελικά για τους πολίτες. Δείχνει ότι η Επιτροπή μας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Για τα πράγματα δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε. Θα ήθελε λοιπόν να μας συμβουλεύσει ο Πρόεδρος. Τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Προς το παρόν, ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε το εξής. Να βρούμε μια διαδικαστική λύση να μην αποφασίσουμε ποιος έχει δίκο και ποιος έχει άδικο στο θέμα Ισραήλ-Παλαιστίνη, να μην μπούμε σε αυτό το ζήτημα, αλλά να εκδώσουμε ένα σύντομο ψήφισμα στην Ολομέλεια βάσει του κανονισμού εργασίας και θα πρότεινα να υποβάλουμε λοιπόν εκ μέρους της Επιτροπής ένα σύντομο ψήφισμα που να αναφέρει την καθυστέρηση, την ουσία της αναφοράς και να ζητήσει από την Ολομέλεια να σχολιάσει και να εγκρίνει, να προτείνει κάποιον τρόπο να προχωρήσουμε. Τουλάχιστον να δείξουμε τι κάτι κάνουμε εμείς σαν Επιτροπή Αναφορών για αυτή την αναφορά. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε το ζήτημα τον Ιούλιο του 2009 προωθώντας το στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων. Και πάλι σαν ήρθε το μπαλάκι πίσω, όπως βλέπετε σε εμά, σχεδόν μετά από δύο χρόνια. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει η κυρία Όκεν. Είχαμε δύο αναφορές, πολύ σοβαρές, μαζί. Δεν είναι θέμα αυτό της ΑΦΕΤ, διότι εδώ έχουμε νομικό ζήτημα ούτε πρόκειται για μποϊκοτάς του Ισραήλ κλπ. Είναι νομικό ζήτημα. Είχαμε καταρχάς μία αναφορά για τη συμφωνία, την σύνδεση, την εταιρική συμφωνία. Και πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στο Ισραήλ, το οποίο είναι μία σύγχρονη πολιτισμένη δημοκρατία, άρα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Πρέπει λοιπόν να τους πούμε ότι ακούστε εδώ, δεν σέβεστε τα κριτήρια συμμετοχής ε, σε αυτή την ε, συμφωνία εταίρων. Άρα λοιπόν παραβιάζετε τη συμφωνία και πρέπει να διορθώσετε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τους χειριστούμε ε, σαν μια σύγχρονη βιομηχανία δημοκρατία, συγγνώμη, να του μεταχειριστούμε έτσι και να του πούμε είσαστε δημοκρατία πολιτισμένη και παραβιάζετε τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας. Ε, όσον αφορά τους οικισμούς, αυτούς που χτίζει το Ισραήλ, δεν μπορούν οι πολίτες του Ισραήλ που ζουν στις, ε, στους οικισμούς αυτούς να τους μεταχειριστούμε ως πολίτες που εμπίπτουν στα κριτήρια αυτής της συμφωνίας. Διότι οι οικισμοί αυτοί είναι παράνομοι και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτούς τους οικισμούς δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νόμιμα προϊόντα της εμπορικής συμφωνίας. Μήπως μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να τους πούμε ότι τα προϊόντα αυτά που έχουν χτιστεί παράνομα σε κατεχόμενο έδαφος δεν μπορούμε εμείς να τα εισάγουμε. Μου έχουν πει ότι 75% των Ισραηλινών προϊόντων που εισάγονται στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από τους παράνομους οικισμούς. Άρα λοιπόν, ίσως εδώ παρουσιάζεται μια λύση και αν σου πούμε παράνομοι οικισμοί και τα προϊόντα από αυτές τις περιοχές είναι παράνομα. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε ε, μέσα στην εμπορική συμφωνία. Λόγια έχουμε πει εκατομμύρια, τώρα πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ. Ε, πολύ σύντομα η κυρία Γκρουνή ναι κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πριν να αποφασίσουμε. Και όσον αφορά την ε, Ολομέλεια, θα πρέπει να συζητηθεί σε... από τους συντονιστές. Άρα, καμία απόφαση σήμερα και θα επιδιώξουμε την αρρωγή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και θα αποφασίσουμε μετά πρόεδρος. Όπως και να έχει, η κυρία Άουκεν ζήτησε να ζητηθεί το θέμα για το Ισραήλ από τους συντονιστές. Επομένως, σήμερα το πρωί τα είπαμε ως συντονιστές, διότι θα πρέπει επομένως στα πλαίσια του προβληματισμού μας, να εκμεταλλευτούμε το ότι σας ενδιαφέρει το θέμα και να το εκπληρώσουμε έτσι άουκεν. Ακόμα και αν η ΑΦΕΤ δεν μας βοηθήσει, θα πρέπει εμείς να το διεκπαιρεώσουμε, γιατί δεν είναι θέμα εξωτερικών υποθέσεων. Είναι θέμα που αποτελεί το θεμέλιο, τη νομική βάση των εργασιών μας. Ναι, κύριε Κλινή, το, το είπε, να το συζητήσουμε και ο συντονιστές ο αναφέρον, ο κύριος Πέγγ ζητεί το λόγο για να το ολοκληρώσουμε και να πάμε στο επόμενο, στο επόμενο που αφορά την δήλωση, την αναφορά, τη δήλωση του κυρίου Χάστινης. Ευχαριστώ. Θα συνοψίσω τι λέμε. Πρόκειται περί νομικού επιχειρήματο. Δεν έχει σχέση με μποϊκοτάζ ή κάποια πολιτική δράση. Πρόκειται περί νομικού επιχειρήματο. Ποιο είναι το γεγονό ότι οι επικισμοί αυτοί των Ισραηλινών σε Παλαιστινιακέ γηέ παράγουν διάφορα αγαθά τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να εισαχθούν στην Ευρώπη. Οπότε συμμετέχει στο εμπόριο αγαθών που έχουν παραχθεί σε παράνομα μέρη επιγεών που εκλάπησαν από κόσμο που έχασε τα πιο βασικά του ανθρώπινα δικαιώματα από πλευρά του Ισραήλ. Κάνοντα το αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομιμοποιεί αυτή, αυτόν τον επικισμό της Παλαιστίνης, συμβάλλει στην ε, παράταση της παρανόμου κατοχής και ε, οδηγεί στην αύξηση των παρανόμων αυτών επικισμών. Αυτά τα προϊόντα είναι παράνομα, τελείω και παύλα. Δεν θα έπρεπε ως ε, κοινότητα ε, να έχουμε συναλλαγές εμπορικές ε, πάνω σε αυτά τα αγαθά. Ευχαριστώ. Κύριε Τάξης, βρίσκεται πάρα πολύ Παντός στο επόμενο σημείο που είναι το υπαριθμόν 12. Ε, θα κάνουμε αυτό το μικρό άλμα, να πάμε από το 9 στο 12 και να τη δουλειά του κύριου Χάστινγκς. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Η επιτυχία τη γνωμοδότησης για πρόσβαση στα έγγραφα Κοινοβουλίου Συμβουλίου και Καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε. Ε, dear President. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να μιλήσω σήμερα όσον αφορά την μεταρρύθμιση του κανονισμού 1049 του 2001 όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα και πιο συγκεκριμένα σχετικά με το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που προετοιμάστηκε από την κυρία Χάνκης. Τον Ιούνιο του 2010, 29 Ιουνίου, ενεστώτος έτους, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέληξε σε μια απόφαση που αναμενόταν πάρα πολύ στην περίπτωση της μπύρας, της βαβαρικής μπύρας. Και εδώ είδαμε πώς μπορεί να προστατευτούν τα, τα, τα δεδομένα και απ' την άλλη να έχει πρόσβαση το κοινό σε έγγραφα, να συμφιλειωθούν τα δύο. Ποια ήταν η λογική που ακολούθησε το δικαστήριο. Ερμήνε τα πράγματα διαφορετικό τρόπο από τον οποίο είχε ακολουθήσει η DPS και εγώ κατά το παρελθόν. Δηλαδή τώρα εργαζόμεθα επί αναθεωρημένου εγγράφου το οποίο θα συμπληρώνει το έγγραφο που είναι στην σελίδα και ένα έγγραφο που δίνει κατευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά τα θεσμικά όργανα και φορεί Ευρωπαϊκή Ενώσεω σχετικά με τη διαφάνεια. Ταυτόχρονα όμω θα γίνονται σεβαστοί κανόνε για την προστασία των δεδομένων και θα δημοσιευθεί το έγγραφο αυτό που ανέφερα πριν το τέλο του έτου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να τονίσω κάτι, ότι η απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την Bavarian Liker για την μπύρα αρκούσε για να ρυθμιστεί αυτή η υπόθεση. Όμως παρέμειναν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και δεν δόθηκε ουσιαστικός προσανατολισμός σχετικά με το πώς οι φορείς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην πράξη. Υπό το φως ε, της αποφάσεως αυτής για τη βαβαρική μπύρα πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ ανοίγματο από τη μία πλευρά και προστασία των δεδομένων από την άλλη πλευρά. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο αν τα θεσμικά όργανα κινηθούν ενεργά, ακολουθήσουν ενεργό προσέγγιση όσον αφορά το θέμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ανάγκη που υπάρχει για άνοιγμα σε ένα πρώιμο στάδιο και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τη σπάση πριν ή τουλάχιστον τη στιγμή που συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, κατά πόσο τα δεδομένα αυτά θα αποκαλυφθούν δημοσία ή δύναται να αποκαλυφθούν. Αυτό συνεπάγεται ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αποφασίσουν όσον αφορά την αποκάλυψη στο κοινό των προσωπικών δεδομένων εκ των προτέρων. Και όχι μόνο μετά που θα ζητηθεί ε, μία πρόσβαση, να ζητηθεί πρόσβαση από κάποιον βάσει τη σχετικη νομοθεσια μια προσεκτική ανάλυση των κανόνων για προστασία των δεδομένων σε άλλο κανονισμό τον 45 του 2001, το 425 του 2001, δείχνει ότι η αποκάλυψη, η υποκάλυψη των δεδομένων καλύπτει ευρύτερο πεδίο από ό,τι υποθέτουν περισσότεροι. Και ακόμα περισσότερο αν το θέμα αυτό αναλύεται σε ένα, τίθεται σε πρώιμο στάδιο. Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων δημοσία επιτρέπεται αν αυτό αποτελεί ένα ανάλογο μέτρο. Αυτό υπογραμμίστηκε ήδη σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σημαντική απόφαση που έλαβε σήμερα το πρωί στην υπόθεση Φόλκερ και Μάρκου Σέλκε που αφορούσε τη δημοσίευση ονόματα δικαιούχων γεωργικών πόρων και τόνισε το δικαστήριο ότι μια σωστή ισορροπία θα πρέπει να επιτευχθεί. Ισορροπία μεταξύ των δημοσίων και των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό πετύει ανάλυση όλων των περιστάσεων μια συγκεκριμένη ε, υποθέσεως. Όμως, όπω βλέπουμε από τη συζήτηση την αναθεώρηση του κανονισμού 1049 του 2001 μέχρι τώρα, υπάρχει όλο και αυξανόμενη συμφωνία που συμφωνεί με την αποφάση του δικαστηρίου, συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου ότι σε, σε πολλές περιπτώσεις μία σωστή ισορροπία ευνοεί την αποκάλυψη των στοιχείων. Αν, παραδείγματο χάρη, τα στοιχεία αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του ατόμου, του ενδιαφερομένου. Το όνομα ενό εμπειρογνώμονα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα, παραδείγματο χάρη, τη έρευνά του ή τη έρευνά τη και τα στοιχεία σχετίζονται αποκλειστικά με ένα δημόσιο άτομο, δημόσιο πρόσωπο που ε, κινείται στα πλαίσια των δημοσίων ιδιωτήτων του. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να δεχτούν μια μεγαλύτερη, μεγαλύτερο έλεγχο από το κοινό όταν κινούνται βάσει της δημόσιας ιδιότητάς του, σύμφωνα με την ομολογία του Λουξεμβούργου και του Σασβούργου Και αν έχουν δημοσιευτεί και τα δεδομένα με σύμφωνη γνώμη του ατόμου, παραδείγματο χάρη σε ένα blog στο διαδίκτυο και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κατά την άποψή μου να μην αποκαλύπτουν τα στοιχεία αν σε ειδικέ περιστάσει, συγκεκριμένε περιστάσει, αυτή η αποκάλυψη θα επηρεάζει αρνητικά τον ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερομένου ή άλλα άτομα που σχετίζονται με αυτόν ή εκείνη. Θα πρέπει ο εμπλεκόμενο να μπορεί να δίνει την άποψή του, να εκφράσει την άποψή του ε, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και ενημερώνει του αρμονισφορεί. Αυτέ οι γενικέ γραμμέ θα πρέπει να κατευθύνουν την ενεργό προσέγγιση ακολουθούν τα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα και οι θεσμοί ε, υπέχουν υποχρέωση να ακολουθήσουν ενεργό προσέγγιση. Αυτό είναι κάτι που απορρέει από την υποχρέωση για ανοιχτή προσέγγιση, είναι υποχρέωση για τη σωστή διακυβέρνηση και σωστή προσέγγιση δυνάμει το άρθρο 1 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως και 15 για την Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και 42, άρθρο 42 τη χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η υποχρέωση για θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν μια ενεργό προσέγγιση επίση είναι κάτι που υπογραμμίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε μια ομιλία στη δική σα επιτροπή στι 29 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια τη συζητήση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία. Και πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα θα κάνουν ό,τι μπορούν, τόσο ώστε να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση, και συζητούμε τώρα το θέμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να δούμε πώς αυτή η υποχρέωση μπορεί να εφαρμοστεί με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όμως, μία ενεργός προσέγγιση δεν μπορεί να επιβληθεί εύκολα από τους πολίτες. Ε, άρα θα πρέπει να συμπληρώνεται μέσω ενός δικαιώματος που έχουν οι πολίτες να ε, υποχρεώσουν εφαρμόζεται η δημόσια πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία και όταν συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικά στοιχεία όταν είναι δίκαιη με τέτοια πρόσβαση. Ένα το δικαίωμα μπορεί να βρεθεί στο σχετικό κανονισμό για την πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία. Με την ερμηνεία που έδωσε το δικαστήριο στην περίπτωση Bavarian Lager, η εφαρμογή του δικαιώματος της του κοινού στα, στη, στα βάση δεδομένου που περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία φαίνεται ότι είναι περιορισμένο και εν πάση περιπτώσει υπόκειται σε όρους που στην πράξη ίσως να είναι δύσκολο να πληρωθούν. Εάν το διαφερόμενο θεσμικό όργανο δεν έχει, αναφε... δεν έχει αποκαλύψει ενεργά αυτά τα στοιχεία και κάποιο θέλει πρόσβαση, εκείνο ή εκείνη θα πρέπει να δώσουν μια δικαιολογία θεμητή ή να προβάλλουν επιχειρήματα που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητα αποκάλυψης αυτών των προσωπικών δεδομένων. Και οι γενικές αρχές για τη διαφάνεια δεν φαίνεται να αρκούν και γι' αυτό το λόγο σε μια πρώτη αντίδραση τον Ιούνιο είχα δηλώσει ότι η απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία και το, λόγο, και το ρόλο που έχει ο νομοθέτης που θα πρέπει να παρέχει πιο σημαντικό, πιο ουσιαστική κατεύθυνση όσον αφορά τα θέματα αυτά. Θεωρώ κρισίμου σημασία λοιπόν να τροποποιηθεί ο κανονισμός 1049 του 2001 ούτω ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί αλλά η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών θα αντικατοπτρίζει μια θεμητή σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του κοινού και του ατόμου. Για τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, αυτές που προανέφερα, με στοιχεία που αφορούν, αφορούν μόνο την επαγγελματική δραστηριότητα του εμπλεκομένου ή ενός δημοσίου προσώπου που δρά στα πλαίσια της δημόσιας ιδιότητάς του ή τα δεδομένα με τη σύμφωνη γνώμη του ατόμου έχουν ήδη δημοσιευτεί, τότε δεν πρέπει να υπάρχει ανάγκη να δίδονται συγκεκριμένοι, να προβάλλονται συγκεκριμένοι λόγοι. Συνεπώ, μετά από την απόφαση για την βαβαρική μπύρα ε, υπάρχουν ακόμα πιο ισχυροί λόγοι για την τροποποίηση του κανονισμού επ' αυτού. Η τροποποίηση επ' αυτού του σημείου που υπέβαλε το Κοινοβούλιο στην, σε 11 ε, Μαρτίου του 2009 στην Ολομέλεια ακριβώς αυτό έκανε. Έδινε σαφείς προσανατολισμούς τεκμηριωμένου και επέτρεπε στον πολίτη τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσει πρώτου δικαστηρίου ή του διαμεσολαβητή ότι η άρνηση αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων δεν αντικατόπτριζε τη σωστή ισορροπία μεταξύ δημόσιου συμφέροντος και ατομικού συμφέροντος. Η αρνηση αποκαλυψη προσωπικων δεδομενων δεν εκθέσεως δημοσιου συμφεροντο και ατομικου συμφεροντος η σχεδιο τη επιτροπη ελευθεριων της 12 η Μαΐου του 2010 επιβεβαίωσε αυτή την τροπολογία, την παγίωσε όπω γνωρίζετε, είναι τροπολογία επαριθμό 44. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η τροπολογία που προτάθηκε ε, όσον αφορά το σχέδιο νομοδοτήσεως της ε, Επιτροπής σας και η τελευταία εκδοχή αυτής που είδαμε ήταν του Ιουλίου του 2010 και είναι η τροπολογία 7 που αφορά το θέμα αυτό, αποτελεί βελτίωση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμφισβήτητα. Όμως δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη σωστή ισορροπία μεταξύ της απέτηση για διαφάνεια και των ιδιωτικών συμφερόντων του εμπλεκομένου. Λοιπόν, εγώ θα συνέστηνα στην Επιτροπή Αναφορών ένθερμα να υποστηρίξει την τροπολογία της εκθέσεως της Ολομελίας της 11 η Μαρτίου του 2009 επ' αυτού, όπως υπευλήθη εκ νέου την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών στην έκθεσή της της 12 η Μαΐου του έτους. Βεβαίως, είμαι στη διάθεση ε, στη διάθεσή σας, αν έχετε ερωτήσεις να απαντήσω οποιαδήποτε στιγμή μετά τη συνάντηση αυτή και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα μπορέσω να σας μοιράσω επίσης το έγγραφο το οποίο σχολίασα και αυτά που είπα για να τα μοιραστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε και ο Πίστερ Χάστινγκ στη δήλωσή του. Δεν ξέρω αν κάποιοι συναδέλφους ε, θέλουν να σχολιάσουν, να υποβάλουν ερωτήσεις ή θέλουν να πούν κάτι για το θέμα. Η κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Χάστινγκ που ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας η συνάδελφος δεν μπόρεσε να προσέλθει, αλλά ξέρετε, είναι η συγκεντριά μας για το θέμα της προσβασιμότητα στα έγγραφα. Πάντως όλα όσα μας είπατε θα τα διαβάσω και έχω να σας ζητήσω μία μικρή διευκρίνηση όσον αφορά την υπόθεση της βαβαρικής ε, μπύρας, γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αντίφαση σχέση με την επιταγή της διαφάνειας που μας εξηγήσατε. Δεν θα πρέπει να δοθεί ένας πιο ξεκαθαρός ορισμός του σχετικά με το τι πάει να πει δεδομένο και τι πάει να πει έγγραφο. Τι είναι δημόσιο, τι είναι ιδιωτικό, άρα να γίνει κάποιο είδου τροποποίηση του σχετικού εγγράφου. Χάστινγκς. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψατε μου να σας τα απαντήσω ή στα αγγλικά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει διερμηνία, έτσι. Οπότε αυτό θα μου βοηθούσε. Λοιπόν, το θέμα του ορισμού του εγγράφου αποτελεί επίσης ένα τμήμα της αναθεωρήσεως και γνωρίζω ότι ο διαμεσολαβητής μεταξύ άλλων επέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το νέο ορισμό, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει κίνδυνος μειώσεως του πεδίου εφαρμογής ε, όλου του κανονισμού, εγώ δεν ξέρω, συμφωνώ με την επίκριση, δεν χρειάζεται να ορίσουμε εκ νέου το έγγραφο για να καλύψουμε το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προσωπικά δεδομένα σε ένα έγγραφο. Δεύτερον, το δικαστήριο, το ευρωπαϊκό, σαφώς δήλωσε στην παρούσα εξαίρεση όσον αφορά το θέμα ότι αυτό συνεπάγεται πλήρη αναφορά στον κανονισμό περιπροστασίας δεδομένων. Αυτό από μια πρώτη ματιά θα έπρεπε να είναι πηγή χαράς για τον Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι στην πράξη αυτό οδηγεί σε περιπλοκότατη ανάλυση πολλών ζητημάτων από πλευρά του ετούντο. Όλα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολύ λεπτόμερο. Και μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι ότι ο αναφέρον θα πρέπει να αποδείξει, ο ετών μάλλον γιατί χρειάζεται τι πληροφορίες. Και αυτό στην πράξη δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα, απαιτεί πολλή δουλειά και πιθανότατα θα οδηγήσει σε δυσανάλογα αποτελέσματα εις βάρος της σωστής ισορροπίας που απαιτείται. Και όπως προανέφερα, το δικαστήριο έλαβε σαφή απόφαση, αλλά δεν έδωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα επιτευθεί ο δύσκολος στόχος. Ο κανονισμός προστασίας των δεδομένων έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να παρέχει λύσεις για διαθροτικές ε, ε, καταστάσεις. Και αυτή η γενική, το γενικό πλαίσιο δημιουργεί πρόβλημα σε λίγες περιπτώσεις στο τέλος. Αλλά δεν δίδεται απάντηση όσον αφορά την ισορροπημένη λύση που απαιτείται για την πρόσφαση του κοινού στα δεδομένα. Εγώ είμαι υπέρ πλέον ουσιαστικών μέτρων, πλέον ουσιαστικών κατευθυνσίων πρέπει να δοθούν. Ευχαριστώ κύριε Hastings. Έχετε κάτι άλλο να πείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας στην Επιτροπή Εναφορών και ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Να συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε, δηλαδή στο σημείο 10. Προέρχεται αυτή η αναφορά από τον Γιώρης Ντεν Μπλάνκεν. Δεν λέει, αλλά φαντάζομαι ότι είναι Ολλανδικής ηθαγενείας. Αν και βέβαια ποτέ δεν ξέρει κανείς και έχουμε επίσης 17 που έχουν προσυπογράψει. Πρόκειται για εξορρυκτικό έργο στο το μισλάβιτσε της Πολωνίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, μεγάλη μας τιμή που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Η Greenpeace είναι μια παγκόσμια οργάνωση προσβέτων των περιβάλλων και στα πλαίσια της πρόθεσης ε, παγκοσμίων λύσεων και καταπολέμησης τη ε, μόλυνση του περιβάλλοντο αντιμετωπίζουν γενικότερη σημασία και αντίκτυπο. Ένα ε, από αυτά είναι και το εξορρυκτικό έργο στο το Μισλαβίτσε της Πολωνίας και θέλω να δώσω το λόγο στον Ηβα Βίος της Greenpeace Πολωνίας ο οποίος θα μιλήσει εκ μέρους όλων εκείνων που υπέγραψαν την αναφορά σχετικά με το εξορρυκτικό έργο του Τομισλαβίτσε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ και να μιλήσω σήμερα. Η αναφορά καλύπτει ευρύ φάσμα οικολογικών, πολιτισμικών και οικονομικών προβλημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στην Πολωνία από ένα εξορυχτικό έργο ε, λιγνίτη στην Τόμισλαβίτσε. Εγώ αναμίχθηκα στο κίνημα κατά το ρηχείο το 2008, έκτοτε συναντήθηκα με, με, τον δήμαρχο της πιο κοντινής πόλης, πολλούς αγρότες και πολλές οικογένειες και πολλούς επιστήμονες που όλοι από κοινού διαμαρτυρήθηκαν κατά αυτού του έργου. Επίσης είδα πώς η περιοχή και οι κάτοικοι της περιοχής επηρεάστηκαν και από άλλα εξορρυκτικά προγράμματα της περιοχής αλλά πολλά μπορούν να διασωθούν για όλο αυτόν τον κόσμο αν μιλήσουν όλοι μια φωνή γιατί αν μιλήσουν μια φωνή και πολεμούν κατά το ξορυχτικό έργο, σημαίνει ότι ε, πολεμάνε για την πατρίδα του, για την πολιτιστική αξία. Ένα τέτοιο κοινό ε, κίνημα αναμειγνύει την κοινωνία των πολιτών που πολεμά για ευρωπαϊκέ αξίε και για νόμου. Πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε να διασώσουμε πολύτιμο, πολύτιμη φυσική ομορφιά τη λίμνη Γκόπο στην Πολωνία που ήταν, ε, είναι βιότοπος για πολλά προστατευόμενα και κινδυνεύοντα είδη. Η λίμνη Γκόπο έχει μεγάλη οικολογική σημασία και έχει σημαντική θέση στην πολωνική ιστορία και στον πολιτισμό της Πολωνίας. Σήμερα στις ακτές της λίμνης μπορεί να πάει σε πύργο μεσαιωνικό που είναι ρήπιο του Καζιμίρ του Μέγα, Πολωνού Βασιλέα. Η πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον τη Πολωνία κινδυνεύει να δημιουργηθεί αυτό το ρηχείο λιγνίτη κοντά στη λίμνη. Πολλοί και οι ντόπιοι δήμαρχοι και επιστήμονε δύο πανεπιστημίων και μη κυβερνικέ οργανώσει πολιτιστική κληρονομιά και απλοί πολίτε και αγρότε διαμαρτυρήθηκαν κατά του ορυχείου το Μισλαβίτσα τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, έχουμε προβάλει επιστημονικά επιχειρήματα, αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου για το ρηχείο και νομικά έχουμε προσφύγει και έχουμε προσεγγίσει και μέλη ε, του Κοινοβουλίου μας με τις ανησυχίες. Παράλληλες προσπάθειες οι Κεντρικέ αρχέ τη Δημοκρατία, τη Πολωνία αποφάσισαν να δώσουν την άδεια για τη δημιουργία του ρηχείου αγνώντας τις προειδοποίησεις ε, των επιστημόνων για τι καταστροφικέ συνέπειε για τη λίμνη Γκόπου και ε, γενικέ αρνητικέ συνέπειες στην περιοχή. Ε, το πρόγραμμα αυτό της Τομισλαβίτσε απειλεί την λίμνη Γκόπο διότι θα δημιουργήσει εκροή υδάτων και θα επηρεαστεί επίσης και την ποιότητα των υδάτων του οικοσυστήματος. Ήδη πολλά ορυχεία στην περιοχή είχαν συνέπειε και είχαν καταστροφικέ συνέπειε. Πολλέ λίμνε έχασαν ακόμα και το 1 τρίτο του, των υδάτων του. Κατά συνέπεια, όχι μόνο η φύση, αλλά και η γεωργία, η αλληλεία, ο τουρισμό και η οικονομική ευμάρεια του λαού τη περιοχή ε, επηρεάζονται. Η κλίμακα τη οικολογική και κοινωνική καταστροφή αναφέρθηκε εκτενώ από τα πολωνικά μέσα ενημέρωση. Εν τέλει, ο λιγνίτη από το ρηχείο όταν κα, καεί σε μονάδε παραγωγή ενέργεια περίπου 50 εκατομμύρια τόνου διοξιδίου του άνθρακο θα εκπέμψει στην ατμόσφαιρα. Ε, καλωσορίζουμε το ότι πεσήμανε την παραβίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο ότι έγινε παράβαση από την Πολωνία. Εδώ παραβιάστηκαν αρκετά άθρα τη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους βιοτόπους και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επίση παραβιάστηκε. Παρά, παρόλα αυτά η πολωνική κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποίησεις και προχωρά στην κατασκευή του ορυχείου. Οι δικαστικές διεργασίες αργούν και ίσως τελικά το έργο να σταματήσει όταν έχουν γίνει επενδύσεις, έχει γίνει το έργο και όταν ήδη είναι, έχουν προξενηθεί ανεπιστευτεί ζημίες. Αντιμετωπίζει πολλές, ε, πολλά προβλήματα η πολωνική οικονομία για την ενέργεια. Η παραγωγή ενέργειας εξαρτάται από τον άνθρακα και το λιγνίτη. Θέλουμε να ξεχρονιστεί ε, το σύστημα ενέργειας να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ξεπεράσει τον άνθρακα η Πολωνία. Ε, το, το έργο της Ομισλαβίτσε δείχνει ότι κάνει ε, λάθος επιλογής η Πολωνία. Βασίζεται στο λιγνίτη και στον άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ε, και δημιουργεί μονοπόλια στην αγορά και δεν ε, δημιουργεί ένα καθαρό σύστημα ενεργειακό και δεν σέβεται το, το περιβάλλον και τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δώσουν μια απάντηση στο θέμα. Σα ζητούμε να επιμείνετε και να πιέσετε τι πολωνικέ αρχέ να σεβαστούν τον νόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράσει κατά παραβιάσεων που συμβιώνται, ώστε το πρόγραμμα τη στο Μισλαβίτσε να σταματήσει πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και θα ήθελα να δηλώσω ότι όλοι σα είσαστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφτείτε αυτέ τι περιοχέ που κινδυνεύουν και την πολύτιμη λίμνη Γκόπο, αυτή καθεαυτή και να συναντηθείτε με του γενναίου εκείνους ανθρώπους που αντιστέκονται σε αυτό το επικίνδυνο και καταστροφικό εξο, έργο. Ευχαριστώ. η κυρία Κοσλόσκα έχει το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα-πρώτα, επιτρέψτε μου να σα τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντηση που καλύπτει τα ζητήματα που αναγύπτουν από την αναφορά περιορίζεται στα του έργου καθ' αυτού. Δηλαδή, επιβάλλεται να γίνει ένα σε αυτού του κλάδου στην Πολωνία. Και όμω και εμεί ασχολούμαστε με τα του έργου ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μα. Επίση, ε, αναφέρθηκε από τον αναφέροντα ότι είχε υπάρξει μια καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί τη βάση της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέβασε μια σειρά επιστολών και διευκρίνιζε το, το τι συμβαίνει σε σχέση με τις ε, πολωνικές αρχές. Και επί τη βάση των ε, πληροφοριών μα παρέσχει η Πολωνία και τη σχετική ανάλυση δεν ικανοποιηθήκαμε. Ότι δηλαδή είχε γίνει μια άρτια αξιολόγηση που έλαβε υπόψη τα όσα επιτάσσουν οι διατάξεις συγκεκριμένα το άρθρο 6 τη, της ε, οδηγίας για το φυσικό περιβάλλον της οδηγίας 42. Οπότε, τον Ιούνιο απευθυνθήκαμε και πάλι στην, ε, στις πολωνικές αρχές και στείλαμε μια επιστολή στην οποία επισήμως επισημάναμε τις διαπιστώσεις μας. Τέλος Αυγούστου, 25 Αυγούστου, ελάβαμε τις σχετικές απαντήσεις. Επίσης είχαμε και αρκετή ε, τεκμηρίωση όσον αφορά τα όσα είχαν να μας πούν οι πολωνικές αρχές για όλα αυτά που αφορούσαν την υπόθεση της ε, αναφοράς. Και γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα που υπάρχει, το πόσο ε, έχει προβληματιστεί ο κόσμος εκεί και βεβαίως θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε την Επιτροπή σας αλλά εν γέννη όλους ότι όταν υπάρχει ε, αυτή η, αυτή η, αυτή η επίσημη επιστολή όπου επισημαίνουμε τις διαπιστώσεις μας τα πράγματα ε, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Δεν ξέρω τώρα αν ο αναφέρον θέλει να υποβάλει επιπλέον ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, ζήτηκαν διευκρινήσεις από την πολωνική κυβέρνηση. Και επομένως, ίσως πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να περιμένουμε και τη νέα απάντηση των Πολωνών. Θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, δύο λόγια. Να μείνει, λέει η κυρία Άουκεν, ανοιχτή αναφορά. Και θα ήθελα επίσης να μάθω τι ισχύει Μήπως θα πρέπει να πάψει η χρηματοδότηση αφού τώρα ομονοούμε. Μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει να δίνει όλα αυτά τα τόσα τόσα τόσα υψηλά κονδύλια για κάτι που θα μπορούσε να γίνει αλλιώς με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φυσικά αυτέ οι κρατικέ επιδοτήσει είναι ένα μόνο μικρό κομμάτι του όλου παζλ. Ένα λεπτό ο αναφέρον και ένα λεπτό η Κομισιόν. Θα είμαι σύντομη, γιατί δεν έχουν υπόψη μα κατά πόσον όντω υπάρχει κάποιο κρατική επιχορήγηση για αυτό το έργο. βεβαίω. και ενισχύεται. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Ο αναφέρον. Ευχαριστώ. Όλο το έργο αυτό είναι κρατικό. Ολόκληρο το έργο. Ε, είναι μια προσπάθεια να, να χτιστεί αυτό το ανοιχτό ορυχείο, το, το ορυχείο επιφανείας από το κράτος. Και ενδεχομένω να μπορεί να δοθεί και εξωτερική ενίσχυση σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το έργο. Γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Σας ευχαριστώ για, αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Αναμένουμε την απάντηση της πολωνικής κυβέρνησης και θα έχουμε μια επόμενη ευκαιρία συζήτησης. Ευχαριστώ. Το 11 είναι από την κυρία Νίβε Σιμπέας Γουέλτα, ε, όνομα 4, ε, αριθμός 428-061 και αφορά την εκτροπή των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Εύρου στους ποταμούς Τέρ και Γιόμπρεγκάτ. Υπάρχει η ετούσα εδώ, είναι εδώ. Όχι, ο Μιγγέλ λοιπόν. Υπήρχε μια σύγχυση με το όνομά σα, είναι ο κύριος Μαρτίνες, συγγνώμη. Ο κύριος Μαρτίνες μιλάει εξ ονόματος της ετούσας. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Αυτή η αναφορά προέρχεται λόγω της ξηρασίας του 2007, η οποία επανήλθε το 2008 και εκδόθηκε ένα βασιλικό διάταγμα για τη διαχείριση της απορροής ε, της, ε, του ποταμού στην Καταλωνία, περιοχή ε, Βαρκελόνης η Ισπανική κεντρική κυβέρνηση σε συνεργασία με την τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας και βάσει του βασιλικού διατάγματος το Απριλίου 2008 αποφάσισε να εκτραπούν τα ύδατα της λεκάνης απορροής στους δύο ποταμούς που αναφέρονται στην αναφορά. Αυτή λοιπόν η απόφαση εκτροπής είναι επίγουσα. Ε, υποτίθεται ότι θα ψηφιζόταν ένας νόμος που θα μας έδινε τη δυνατότητα αξιολόγησης εάν το, η εκτροπή αυτή θα ήταν προσωρινή, ένα προσωρινό έργο ή μία μόνιμη εκτροπή. Τώρα, βλέποντας ε, τα, σχέδια. Πιστεύουμε ότι η εκτροπή αυτή θα είναι μόνιμη και μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι επιπτώσεις αυτής της εκτροπής. Έχουμε βεβαίως ξηρασία, αλλά η ξηρασία δεν διαρκεί για πάντα και γι' αυτό μας ενισχύει η μονιμότητα αυτής της πρόχειρης υποδομής. Και δεν πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει άλλα έργα αφαλάτωσης τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, ούτε έχει γίνει μελέτη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακής χρήσης. Ούτε έχει γίνει διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης των υδάτων των δύο ποταμών. Άρα λοιπόν πολλά κριτήρια και πολλές προϋποθέσεις για την έγκριση της μελέτης δεν έχουν γίνει σεβαστά ούτε οικονομικές επιπτώσεις της μελέτης απορροής των υδάτων. Και τελικά έτσι επιδικάστηκε αυτό το έργο στις 8 Μαΐου. Άρχισε βροχή όμως. Και η καταλανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο, οπότε και στις 6 ε, Ιουνίου η Ισπανική Κεντρική Κυβέρνηση θεώρησε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προς τούτο. Εμείς διαβάσαμε την καταγγελία στην Κομισιόν, που δεν έκανε τίποτα, γιατί θεωρήσαμε ότι εδώ έχουν επικαλεστεί κατάσταση ανάγκης αλλά κάτι το οποίο δεν θεμελιωνόταν και θεωρήσαμε ότι αυτό είναι κάτι που αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. Δεν υπήρχε πονή λοιπόν ίδια αντίδραση από την Κομισιόν όπως από τη δική σας Επιτροπή. Και... Αναβαθμίσαμε, επεκτείναμε την καταγγελία μας όταν υπήρχε και σχετική δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών και ο Επιτρόπος ο κ. Δήμας αναγνώρισε ότι κατόπιν καταγγελία του κ. Ρούχο του Ευρωβουλευτή ότι δεν έχει λάβει κάποια επικοινωνία, κάποια ανακοίνωση από την Ισπανική κυβέρνηση Θεωρήθηκε δε ότι σήμερα το άρθρο 2 της σχετική οδηγίας δεν είχε γίνει η αναγκαία μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, η απόφαση Ισπανικής κυβέρνησης είχε ισχύ νόμου και ούτε αυτό το έγγραφο είχε διαβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θεωρήθηκε επομένως ότι καλυπτόμαστε από την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών. Και έτσι εμείς καλυφθήκαμε. Υπάρχει πρόβλημα. Στις 12.30 θα σταματήσει η διερμηνία, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε παρακαλώ θα πρέπει να ολοκληρώσετε γιατί ήδη έχει ε, ολοκληρωθεί το ωράριο και παίζουμε τις παρατάσεις. Συνεχίζει ο μιλητής. Οπότε και έτσι είδαμε ότι ήταν ε, αυτό ένα δικονομικό τέχνασμα ε, και επομένως δεν θα έπρεπε να εφαρμοστεί ε, αυτό το οποίο είχαν αποφασίσει στην κυβέρνηση. Γιατί ρητός αναφέρεται τα κράτη-μέλη δεν είναι δυνατόν να προβούν σε κάποια μέτρα τα οποία θα θέσουν εν κινδύνο την υλοποίηση της συνθήκης. Και λέτε σε περίπτωση που τυχόν υπάρχει κίνδυνος. Ε, σε υγιείς περίπτωση που τυχόν τεθεί εις εν αμφιβόλο η συνθήκη. Και επομένω ε, το 2002 έχουμε απόφαση τη Κομισιόν σε σχέση με τη βελτίωση τη εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου. Και εκεί πέρα αναφέρονται ρητό κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να σταματούν οι επιζήμιες πράξεις. και γι' αυτό και αναφερόμεθα ή στα σκουπίδια στην εξοχή ή για την, την καταστροφή των δασών για λόγους ε, ανοικοδόμησης. Επόμενος είχαμε πει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κάποιο ασφαλιστικά μέτρα. Δεν έγινε εδώ πέρα τίποτα. Ούτε επίσημη ανακοίνωση διαβάστηκε εκεί που έπρεπε. Ούτε καν στις, στις δημοσιεύσεις εφημερίδες έγιναν εδώ πέρα βάζω τελεία κύριε Πρόεδρε και σε ευχαριστώ. Ο κύριος Χόρχη Ρομέρο όμως τώρα λέει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την αναφορά πρώτα-πρώτα εδώ διαπιστώνεται ότι έχουμε αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμα ενισχύ και επομένω δεν έχει ε, νομικέ συνέπειε και επομένω και εμεί δεν μπορούμε τώρα να αξιολογήσουμε κατά πόσον αυτό το, ε, το, το, το, το, το νομοσχέδιο ε, το, το οποίο έφερε αυτές τις συνέπειες όσον αφορά αυτό το, το έργο είναι κάτι το οποίο είναι σύντονο με το κοινωτικό δίκαιο. Διότι στην αιτιολογική έκθεση αυτό το νομοσχέδιο έλεγε ε, αυτό, αυτό έλεγε ότι ο στόχο είναι να υπάρχουν κάποιε εγγύσει βραχυπρόθεσμε όσον αφορά ε, το, το, να υπάρχει αρκετό νερό για τα 5 εκατομμύρια κατοίκων τη Βαρκελόνη και εξηγείται εις, αυτό το διάταγμα ότι ε, εάν είχαμε τη, τη βροχή αυτή που έγινε ότι θα υπήρχαν προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διορθωθούν μέχρι ότου αρχίσει να τον ε, να λειτουργεί το τον Ιούνιο 2009 αυτό το εργοστάσιο αφαλάτωσε στο, στο, στο Πράντε Λιομπρεγκάτ και εδώ πέρα υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη ρήτρα, η διάταξη όπου διευκρινίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχει λήξει το ωράριο εργασίας των ε, διερμηνών, οπότε τώρα να μας τα πείτε στα αγγλικά για να καταλάβουμε όλοι. I have no problem in speaking in English. You have a problem speaking? No, you don't have any problem, so speak. So continue in English. Yes. And... Okay.